Καλημέρα και να ξεκινήσουμε παρακαλώ τι συνεδριάσει μα και σα καλωσορίζω στην ε, Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Σήμερα το απόγευμα θα κοιτάξουμε λοιπόν την ημερήσια διατάξη. Εγκρίνεται η ημερήσια διατάξη μια και δεν έχω λάβει ε, αιτήματα για αλλαγή τη ημερήσια διατάξη στι ανακοινώσει. Κοιτάξτε παρακαλώ τις γλώσσες ε, οι οποίες διατίθενται. Ελληνικά μπορείτε να ακούσετε και να μιλήσετε και έτσι περνάμε στο τρίτο σημείο της ημερησία Έχουμε σήμερα μία μελέτη την οποία θα παρουσιάσουμε, μία αξιολόγηση της δεκαετούς ε, διαδικασία συνεργασίας και επαλήθευση ε, για την Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Cooperation and Verification Mechanisms και η οποία λαμβάνει χώρα στα πλαίσια τη αρμόδιας γενική γραμματείας. Έχουμε κοιτάξει το θέμα αυτό Επισταμένως έχουμε πλέον κλείσει 10 χρόνια και έχουμε διαπιστώσει ότι θα ήταν σημαντικό πέρα από τις εκτέσεις Προέδρου να κάτσουμε να κοιτάξουμε το θέμα των προόδων που έχουν γίνει συνολικά στην, στις εκτάσεις Προέδρου. Πρώτο, να καλωσορίσω τους υπεύθυνους κατάρτισης της έκθεσης αυτής του CSS, το κέντρο ε, τέτοιων ε, παρουσιάσεων και αναλύσεων. Να τους δώσω το λόγο για να μα παρουσιάσουν την έκθεση του. Πάρα αυτά παρακαλώ να συστηθείτε κιόλα να πείτε δύο λόγια για το τι, ποιοι είστε και τι κάνετε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μα καλέσατε σήμερα το απόγευμα για να σα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα τη μελέτη μα για τη συνεργασία, για το μηχανισμό συνεργασία και επαλήθευση. βουλγαρια Βουλγαρία-Ρουμανία. Και χαιρόμαστε που έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τα χωρίσματα τη έκθεσης. Θα μιλήσουμε 15 λεπτά περίπου και μετά από κάποια εισαγωγικά σχόλια τα οποία θα κάνω εγώ, θα δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου, τον Στέφαν Κρόιτς, ο οποίος και θα μας παρουσιάσει κάποια από τα βασικά πορίσματα για την Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Και στο τέλος θα παρουσιάσω κάποια συνολικά συμπεράσματα για τις δύο χώρες εγώ πάλι. Πολύ ωραία. Να ξεκινήσουμε με τις να κάνουμε μία επανάληψη σε ό,τι αφορά το σκοπό του συγκεκριμένου εγχείρηματο. Τέσσερις ήταν οι στόχοι. Να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος του, του μηχανισμού στις δύο χώρες τα τελευταία δέκα χρόνια και πιο συγκεκριμένα τι πρόοδος έχει σημειωθεί για την επιτεύξη των διαφόρων οροσίμων. Κατά τρίτον, να εξεταστεί η πρόοδο ό,τι αφορά την εφαρμογή των συστάσεων που έγινε από το Συμβούλιο και την Επιτροπή πέρσι στι αρχέ του έτου και τέλο να εξεταστεί ο ίδιος ο μηχανισμός καθεαυτός, πώς λειτουργεί, κατά πόσο να έχει επιφέρει τι αλλαγέ που επιθυμούσαμε. Η έρευνα έγινε σε μία περίοδο μεταξύ του Αυγούστου και του τέλους του Νοεμβρίου του περσινού έτους Έγιναν συζητήσεις και στις δύο χώρες, αλλά έγιναν μάλλον συζητήσεις με 25 άτομα από τις δύο χώρες που εκπροσωπούσαν την κυβέρνηση, τις διάφορες υπηρεσίες, ε, το δικαστικό σώμα, μικείο, εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις χώρες αυτές. Έγιναν επίση συζητήσεις και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση με την Γενική Διεύθυνση Justice Home της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. και όταν ολοκληρώθηκαν οι έρευνε και οι διαβουλεύσει, έγιναν διάφορα εργαστήρια σε κάθε χώρα, στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία για να συζητηθούν τα απορίσματα τα οποία ανέκυπταν ε, εν την παρόδο με τους βασικούς εμπλεκόμενους φορείς ε, να αναφέρω κάποια στοιχεία τώρα για τον, για μηχανισμό, το CVM. Εισήχθη το 2007 ως ένας τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων σε θέματα κράτους δικαίου στις δύο χώρες. Η βάση του μηχανισμού CVM ε, είναι μία σειρά από ορόσημα, από στόχους 6 για τη Βουλγαρία, τέσσερις για τη Ρουμανία σε ό,τι αφορά τη δικαστική μεταρρύθμιση, την καταπολέμηση της διαφθοράς, στην περίπτωση της Βουλγαρίας και σε ό,τι αφορά το οργανωμένο έγκλημα. Διατέθηκε σημαντική χρηματοδότηση, σημαντική πόρη για τη μεταρρύθμιση στις δύο χώρες, 81 εκατομμύρια ως τώρα στη Βουλγαρία και περίπου 150 εκατομμύρια ως τώρα στην Ρουμανία από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο και Ταμείο Επενδύσεων, αλλά και, το... και από το Ταμείο ISIC. E Υποστηρίζονται η χρήση διακυβέρνηση, η βελτίωση στις ε, δημόσιες ε, προμήθειες, στις κτλ. Και έγιναν ε, τεχνικές εκθέσεις πρόοδου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες αξιολογήσεις. Τώρα θα να δώσω το λόγο στον συναδελφό μου, τον Στέφαν Κρόιτς, για να μας παρουσιάσει τα συγκεκριμένα πορίσματα για τη Βουλγαρία και την Ρουμανία και στο τέλος θα, κάνω, θα συνοψίσω πάλι. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση για τη Βουλγαρία. Σημειώνουμε ότι η πρόοδος δεν ήταν όσο ταχεία όσο αναμενόταν πριν από 10 χρόνια όταν συστάθηκε για πρώτη φορά ο μηχανισμός σημειώθηκαν και εξακολουθούν να σημειώνονται βασικές, ε, βασικά ζητήματα σε ό,τι αφορά την αντιμετωπίση της διαφθοράς, της ενίσχυσης του δικαστικού σώματος, στην ανεξαρτησία του και στην καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματος. Παρ' όλα αυτά, ο μηχανισμός CVM μας βοήθησε, βοήθησε τη Βουλγαρία να εστιαστεί σε θέματα μεταρρυθμίσεων και παρά τι συχνέ αλλαγέ κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια, το οποίο προφανώ επιβράδυνε την εφαρμογή διάφορων μεταρρυθμίσεων, σε ό,τι αφορά το οργανωμένο έγκλημα συγκεκριμένα, σημειώθηκε καλή πρόοδο κατά πολέμηση οργανωμένου εγκλήματο, σε ό,τι αφορά την εξαρτησία και τη μεταρρύθμιση του δικαστικού σώματο και εδώ Διαπιστώνουμε ότι πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα και ιδιαίτερω επισημαίνουμε ότι κάποιοι από του εμπλεκόμενου φορεί με τι οποίε έγιναν διαβουλεύσει επισήμαναν διάφορα προβλήματα σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τι αρμοδιότητε και την εξουσία του εισαγγελέα. Επίση, παρακολουθούμε τι αλλαγέ και τι προόδου σε ό,τι αφορά διάφορε περιπτώσει και υποθέσει υψηλού, διαφθορά σε υψηλά επίπεδα. Εδώ διαπιστώνουμε ακόμα προβλήματα και ελλείμματα. Υπάρχει ωστόσο πολιτική θέληση και βούληση της τελευταίας κυβέρνησης να εφαρμόσει τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν από ένα έτος. Ενδεχομένως δε αυτό να πάρει και πιο πολύ χρόνο από ό,τι αναμενόταν πριν από ένα χρόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κοιτώντα τι έγινε στη Ρουμανία, σημειώθηκε σημαντική πρόοδο. και σε ό,τι αφορά και του τέσσερα, τα τέσσερα ορόσημα, του τέσσερις στόχου που είχαν τεθεί για τη Ρουμανία, ιδιαίτερου δε για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού σώματο, όπω και στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία διαπιστώνεται ότι χρειάζονται να ληφθούν πιο πολλά μέτρα για να αποφευχθεί η διαφθορά σε υψηλά επίπεδα και σε τοπικό επίπεδο. Και μια και έχουν γίνει ήδη σημαντικές μεταρρυθμίσει στη Ρουμανία. Τώρα πλέον επικεντρωνόμαστε στη μόνιμη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων αυτών, προκειμένου να δημιουργηθεί και ένα προηγούμενο και πλέον να μην υπάρχει περιθώριο αλλαγή. Αυτό λοιπόν όντω σιγά σιγά επιτυχάνεται. Είμαστε αισιόδοξοι ότι οι συστάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρσι, που ήταν περιορισμένε στον αριθμό, μπορούν να εφαρμοστούν προκειμένου να ολοκληρωθεί ο μηχανισμός CVM για τη Ρουμανία. Και έτσι λοιπόν να διακοπεί. Μεσοπρόθεσμα. Τώρα κοιτώντα τα κοινά ζητήματα που αφορούν και τις δύο χώρες διαπιστώθηκε ότι ο μηχανισμός CVM δίνει σημαντική τεχνική και οικονομική αρρωγή την οποία πραγματικά αξιολογούν και από τις δύο χώρες οι εμπλεκόμενοι φορείς, κάτι που σημειώνουμε. Δεν είναι τεχνική μόνο η διαδικασία αυτή. Η πολιτική βούληση είναι σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία της μεταρρύθμισης, των μεταρρυθμίσεων, της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων. Όχι μόνο να οριστούν αυτοί οι κανόνες, αλλά να υλοποιηθούν πραγματικά. Και έτσι ο μηχανισμός CVM είναι σημαντικός ε, για τη λογοδοσία της εκάστοτε κυβέρνησης και έτσι ενισχύεται η κοινωνία των πολιτών γιατί προστίθεται μια διάσταση εξωτερική, ε, αν θέλετε, εξωτερικού ελέγχου στην όλη διαδικασία σε ό,τι αφορά την έκθεση πρόοδου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύουμε ότι χορηγήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαρκεί πληροφορίε προκειμένου να γίνει αξιολόγηση τη πρόοδου των ε, μεταρρυθμίσεων και τεχνικέ επίση εκθέσει. Δίνουν μια λεπτομερή ανάλυση τη κατάσταση επιτόπου κοιτώντα τώρα τα ορόσημα, τα benchmarks που έχουν οριστεί και για τις δύο χώρες, ασκήθηκε κάποια κριτική ότι ήταν πολύ ασαφή αυτά τα ορόσημα και ότι δεν επέτρεπαν την πραγματική καταμέτρηση της πρόοδου σε ό,τι αφορά δηλαδή το πότε και πώς επιτεύχθηκαν οι στόχοι. Κάποιοι επέκριναν και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι άλλαξε τους στόχους που είχε θέσει στην διάρκεια αυτή της δεκαετούς ε, περίοδου. Δεν προκαλεί ασφαλώ έκπληξη το γεγονό ότι σε μια περίοδο 10 ετών κάποιοι από του στόχου έχουν καταστεί πλέον παροχημένοι. Και είναι δύσκολο να θεωρούμε πότε πλέον οι μεταρρυθμίσεις θεωρούνται μόνιμες. Πότε θεωρούμε ότι έχει επιτευχθεί αυτή η μόνιμότητα. Ιδιαίτερα όταν υπάρχουν αλλαγέ. Ε, μάλλον ένα παράγοντα είναι οι διάφορε αλλαγέ κυβέρνηση και φυσικά ε, η νομολογία σε ό,τι αφορά και το ιστορικό των, κατα... της καταδίκης διάφορων περιπτώσεων και υποθέσεων ε, υψηλή διαφθορά. Θεωρούμε συνολικά ότι ο μηχανισμό CBM είναι χρήσιμο, ωφέλιμο από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρησιμοποιείται για να εφαρμοστεί το κράτο δικαίου στα κράτη-μέλη και σε ό,τι αφορά την άμεση αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων, αλλά και σε ό,τι αφορά τη σωστή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων από πλευρά επενδύσεων δε στι δύο χώρε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουν οι επενδυτέ ότι πραγματικά υπάρχει κράτο δικαίου. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο για να βγάλει τα γενικά συμπεράσματα. Να συνοψίσουμε από αυτά που ακούσαμε. Συμπέρασμα είναι ότι ο μηχανισμό συνεργασία και ελέγχου είναι ένα πλαίσιο πολύ χρήσιμο τόσο ώστε να βοηθήσουμε στις μετερρυθμίσεις δύο αυτές χώρες είναι ένας καταλήτης αλλαγής και θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτά θα γινόντουσαν έτσι κι αλλιώς αλλά θα έπαιρναν πολύ περισσότερο χρόνο οπότε έτσι επιταχύναμε την μεταρρύθμιση και δώσαμε ένα έναυσμα για τις ε, αλλαγές οπότε διαπιστώνουμε πρόοδο σε σχέση με τα κριτήρια αυτά που είχαν τεθεί σε αυτές τις δύο χώρες στη Ρουμανία, την Βουλγαρία και οι δύο χώρες όμως θα πρέπει μέχρι το τέλος της παρούσης θητείας της Κομισιόν να πετύχουν τους στόχους τους πλήρως. Για να δούμε τώρα για το μέλλον. Έχουμε τρεις βασικές επιλογές. Πρώτα-πρώτα όσον αφορά το status quo. Πρώτη επιλογή όσον αφορά τον μηχανισμό όσο έχει σήμερα σε σχέση με τα ορόσημα τα οποία έχουν υλοποιηθεί Άλλη δεύτερη επιλογή είναι να γίνει αλλαγή του μηχανισμού ή να μια όλος διάφορη προσέγγιση. Τώρα σε σχέση με οποιαδήποτε αυτές τις επιλογές δεν θα πρέπει να δούμε τι γίνεται πολύ μακριά στο μέλλον γιατί έχουμε κάποια πρόοδο οπότε θα πρέπει να πιάσουν τόπο αυτές οι βελτιώσεις να δούμε ποιες είναι και οι διαφορές μεταξύ των δύο χωρών, διαφορές προσέγγισης για αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Και επομένως, η δεύτερη επιλογή είναι ένας μηχανισμός παρόμοιος. Ο CVM δηλαδή τροποιημένος ίσως να αλλάξουν αυτά τα benchmark, τα ορόσημα, να έχουμε ίσως κάποιες άλλες ε, προθεσμίες για την υλοποίηση επόμενη τετραετία, ώστε να είναι καλύτερο. Ή να έχουμε έναν άλλον πιο πλήρη μηχανισμό που να καλύπτει και άλλες χώρες, όχι μόνο αυτές τις δύο. Στο Union Pack για δημοκρατία, κράτους δικαίου, ε, δικαιώματα σε σχέση με τον μηχανισμό εκθέσεων της Ένωσης για καταγωγή της διαφθοράς, ίσως στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ε, σε συνδυασμό ίσως και με τον CVM ή ίσως να το συνδυάσουμε με μια ευρύτερη προσέγγιση δηλαδή περισσότερος έλεγχος, περισσότερη αξιολόγηση στα σχετικά μέτρα ε, ε, και συμμόρφωση από τα ίδια τα κράτη-μέλη και να αναλάβουν πιο πρωταγωνιστικό ρόλο οι εθνικές τοπικές αρχές για αξιολόγηση και έλεγχο. Όπως είπε και ο Στέφαν, είναι πολύ σημαντικό για μας, όχι μόνο να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση, αλλά και να ε, παγιωθούν αυτές οι επιτευχθήσεις αλλαγές σαν κάτι το ανέκλητο. Επίσης, όπως φέρθηκε το κλειδί για την επιτυχία το να πιάσουν τόπο αυτές οι αλλαγές και για τα όσα εκκρεμούν είναι υπάρχει πολιτική βούληση προς τούτο. Πολύ σημαντικό αυτό. Και για τις δύο χώρες πάντως, επί τη βάση των ε, όσων διαπιστώσαμε, ε, είμαστε αισιόδοξοι και πάλι σας ευχαριστούμε. Όσο δώσετε την ευκαιρία να σα παρουσιάσουμε τη μελέτη μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και πολύ σημαντικά για μας, γιατί παρακολουθούμε τις ε, εξελίξεις στα δύο κράτη με διαφορετικά επίπεδα ανησυχίας ε, και ενδιαφέροντος βέβαια, με πολύ ενδιαφέρον πάντα. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Μουρομπελκίβου, επικεφαλής στα θέματα της δικαιοσύνης από τη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ρουμανίας και αντίστοιχα τον εκπρόσωπο της Βουλγαρίας για τα ίδια θέματα, κύριε Σαμανστίνκα, από τη μόνιμη αντιπροσωπεία. Τώρα δεν ξέρω ποιος από όλους θα ξεκινήσει, ποιος θέλει να λάβει το λόγο. Παρακαλώ. Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι. Βουλευτές, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι προσκεκλημένοι. Για να ξεκινήσω, θα ήθελα εξ ονόματος των Ρουμανικών Αρχών να ευχαριστήσω αφενός με την Επιτροπή του δημοσιονομικού ελέγχου, του ελέγχου του προπολογισμού για την πρωτοβουλία αυτή που αναλαμβάνει 10 χρόνια μετά την θέση σε εφαρμογή αυτού του κανονισμού και βέβαια και τις υπηρεσίες μελέτης για την ε, ανάλυση και τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς. Θα ήθελα ξεκινώντας λοιπόν να πω ότι είναι αναμφιβολή η χρησιμότητα του μηχανισμού αυτού, επιτρέπει να προχωρήσουμε και να με τις μεταρρυθμίσεις του δικαστικού συστήματος ιδιαίτερο, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ε, ε, χρηστή διαχείριση σε κάθε επίπεδο. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε μια μελέτη πλήρη που καταγράφει τα αποτελέσματα της Ρουμανίας και το γεγονός ότι δεν ε, κινδυνεύει από δρόμο σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό χάρη στην ε, στράτευση των ε, αρχών και σε εθνικό επίπεδο, αλλά και χάρη στην ε, συνεργασία του Ρουμανικού κράτους με τις ευρωπαϊκές αρχές. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να σημειώσουμε ότι και η κοινωνία των πολιτών έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έχει συνεργαστεί σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις. τα κριτήρια της αποφάσεως της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την εκκίνηση του μηχανισμού του 2006 βλέπουμε ότι έχουν οδηγήσει σε μια σαφή πρόοδο. Οι στόχοι όπως καταγράφονται έχουν σε μεγάλο βαθμό έγγραφη ε, στις στρατηγικές της χώρας και τα προγράμματα. Και βέβαια αντιλαμβάνεστε φαντάζομαι τις προσδοκίες των ρουμανικών αρχών σε σχέση με την υλοποίηση αυτών των στόχων. Διαρκώς οι αρχές του Βουκουρεστίου υπογραμμίζουν τη βούλησή τους για πλήρη εφαρμογή των υπόλοιπων κριτηρίων της Επιτροπής του 2017 με τα σημεία αναφοράς που επιδιώκουμε να υλοποιήσουμε ώστε να ολοκληρωθεί αυτός ο μηχανισμός. Περιμένουμε λοιπόν με αδημονία στο πλαίσιο αυτό την προσεχή έκθεση του 2018 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ελπίζουμε ότι θα επιβεβαιώσει πως έχουμε πλήρως επιτύχει τους στόχους για το μηχανισμό συνεργασίας και επαλήθευσης. Μπορώ να πω ότι θα επιτρέψει στη Ρουμανία να βρεθεί στο ίδιο επίπεδο με τα άλλα κράτη δηλαδή οριζόντια εγκάρσια συνεργασία και κάθε τομέα του μηχανισμού. Και πιστεύουμε ότι οι μέθοδοι που ακολουθούμε θα δείξουν ότι μπορούμε να ελοπίσουμε τους στόχους. Ολοκληρώνω έτσι την παρέμβασή μου και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Η Βουλγαρία έχει πει ότι δεν θα συμμετάσχει στο κύκλο, αλλά έχει εκπροσώπους εδώ, αν θέλετε να λάβετε το λόγο. Θέλω να επισημάνω ότι... Παρακαλώ, ναι. Πρόεδρε, στο συγγνώμη. Είναι η πρώτη φορά που λαμβάνω το λόγο, επομένως δεν ήξερα ακριβώς πώς να σας ζητήσω το λόγο. Είναι η πρώτη φορά που είμαι εδώ. Σας ευχαριστώ. Σήμερα ποιος είστε, λέει η Πρόεδρος εκπροσωπώ τη μόνιμη αντιπροσωπεία της Βουλγαρίας. Είμαι μέλος της ε, ομάδας του Μηχανισμού Συνεργασίας και Παλήθευσης. Καλώς ήρθατε, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Ευχαριστώ και τα μέλη της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των κρατών μελών που προσωπούνται εδώ. Είναι μεγάλη χαρά για μας και μεγάλη ευκαιρία να παρακολουθούμε τα ευρήματα αυτής της μελέτης, της έρευνας, που θα διαβιβαστούν βεβαίω στη Σόφια και είμαι βέβαιος ότι θα γίνουν δεκτά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μπορώ να συμφωνήσω με πολλά από τα ευρήματά σας, δηλαδή ο μηχανισμός είχε καταλητικό ρόλο για την εξασφάλιση θετικών αλλαγών στη Βουλγαρία, αλλά και για μια διαδικασία συνεργασίας μεταξύ αρχών και κοινωνίας των πολιτών, αλλά και εξαιρετική συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με χαρά επίσης ακούω πως από την έκθεση καταγράφεται η πρόοδος παραδείγματι για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο, ενό τομέα που έχουμε ήδη πολύ σε επιδόσει, αλλά και για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα. Σα ευεβεβαιώ πω η Βουλγαρία είναι αποφασισμένη να εξασφαλίσει απτά αποτελέσματα για εκείνες ακόμα τι ολίγες συστάσει για τις οποίες καταγράφεται πω χρειάζεται περαιτέρω πρόοδο, δηλαδή η καταπολέμηση τη διαφθόρα και πρόκειται να υιοθετηθεί σύντομα ε, νέο νομοθέτημα που θα εδρεώνει και σε θεσμικό επίπεδο την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Πιο συγκεκριμένα, ως προς την ανάγκη για πιο σαφείς προστοκίες για την Βουλγαρία με βάση τις συστάσεις του Ιανουαρίου του 2017, αλλά και όπως είπε ο Ρουμάνος συνάδελφος, θέλω να επισημάνω και εγώ ότι πρέπει άπαξ και ολοκληρωθεί ο μηχανισμός να βρισκόμαστε σε ίσο πεδίο σε ισότιμο πεδίο συνεργασία με τι υπόλοιπε αρχέ. Η Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ που πήρατε το λόγο. Θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους που ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό. Πρώτα η κυρία, ο κύριος Μπερίνσκι από τη Βουλγαρία. Πυρίνσκι, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να εκδηλώσω την ε, εκτίμησή μου, την δική μου αποτίμηση για τις ε, προόδους, να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους των δύο κρατών για τις παρατηρήσεις και τις τοποθετήσεις τους. Όπως υπόθηκε ήδη, το αντικείμενο του μηχανισμού αυτού συνεργασίας και επαληθεύσης έχει πολύ μεγάλη σημασία και είχε σε όλη αυτή τη δεκαετία πολύ μεγάλη σημασία και αντίκτυπο στη Βουλγαρία και τη, Βουλγαρία, και τη Ρουμανία ασφαλώς. Βλέπω μια ημερομηνία 9 Ιανουαρίου. Δεν ξέρω όμω ε, οι συντάκτε αν ήταν σε θέση να παρακολουθήσουν τι τελευταίε εξέλιξει στη Βουλγαρία, τι σχετικέ με την υπόθεση αυτή. Ο εκπρόσωπο τη μόνιμη αντιπροσωπεία αναφέρθηκε σε ένα νέο νομοθέτημα που προχωρεί προ ολοκλήρωση και εφαρμογή και είναι νόμος ειδικό με στόχο την αντιμετώπιση της διαφθοράς και ειδικότερα της διαφθοράς σε στενότερα κλιμάκια τη κυβέρνηση. κυβέρνησης και βέβαια έχει συστηθεί εντελεχώς και στο Κοινοβούλιο, αλλά και στην κοινωνία της Βουλγαρίας. Ένα από τα πιο φλέγοντα ζητήματα ήταν ο προσδιορισμός ε, της ηγεσία του επικεφαλής αυτού του ε, φορέα η αντιπολίτευση ζητεί να είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ως ανώτατος πολιτικός άρχον, ενώ στην ε, πλειοψηφία του Κοινοβούλου υποστηρίζει την πρόταση που περιέχεται και στο σχέδιο του νόμου επικεφαλής του φορέα να είναι πρόσωπο που θα εκλέγει το Κοινοβούλιο. Την πτυχή αυτή την αναφέρω γιατί θεωρώ πως σε μεγάλο βαθμό έχει να κάνει με τα όσα έχουμε συζητήσει. Το γεγονός ότι δεν είναι τόσο ικανοποιητικά τα αποτελέσματα ως προς την ε, αντιμετώπιση της διαφθοράς. Δηλαδή η νομοθεσία υπάρχει, τα τελευταία χρόνια εισήχθη μια σειρά διαφορετικών αρχών, φορέων που έχουν ως αντικείμενο δράση σε κάποιο τομέα της καταπολέμησης διαφθοράς. Πρόκειται όμως για μια διαδικασία η οποία αν ε, δεν μπορώ να πω παρακολούθηκε ίσως, αλλά πάντως κατέστη δυσχερής λόγω της πολιτικής αντιπαράθεσης. Στο Κοινοβούλιο πριν από μερικές ημέρες ακόμη ε, η αντιπολίτευση σήγαγε ψήφο δυσπιστίας εναντί, έτοιμα δυσπιστίας εναντί της κυβέρνησης επικαλούμενη ζητήματα της διαφθοράς, ότι δηλαδή δεν καταπολεμείται επαρκώς. Δυστυχώς στην κοινωνία το θέμα αυτό έχει πάρει περισσότερο διαστάσεις πολιτικής αντιπαράθεσης, εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης και όχι ως μια προσπάθεια κοινή, με κοινή βούλευση, η βούληση για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Έχω λοιπόν κάποιες ερωτήσεις προς τους συντάκτες της μελέτης για το θέμα αυτό, καθώς ανέφεραν, και είναι σωστό αυτό σε έναν βαθμό, ότι ο ίδιος ο μηχανισμός είχε καταλητική ε, δράση. Διερωτώ με όμως εάν οι συντάκτες ε, θεωρούν ότι έχει μετατραπεί η παραλαμβανόμενη διατύπωση των μελετών και εκθέσεων αν αυτή έχει μετατραπεί σε ένα είδος ρουτίνας, χωρίς το ουσία δηλαδή. Και δεύτερον, διερωτώ με, το Κέντρο για Στρατηγική και Αξιολόγηση. Τι ακριβώς είναι. Έχουν, ε, επί παραδείγματι, ασχοληθεί ε, οι υπηρεσίες αυτές για την στρατηγική και την πολιτική, ειδικά με την καταπολέμηση ευθοράς μόνο, ή μήπως έχουν διαρωτηθεί και αν είναι αυτός ο καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπιση ευθοράς σε χώρες όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία τις έχουν αντιμετωπίσει ως ειδικέ περιπτώσεις ή έχουν ακολουθήσει μια συγκριτική προσέγγιση για αντίστοιχα προβλήματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ασφαλώς σε ένα βαθμό ή σε κάποιους βαθμούς τα ίδια προβλήματα τα αντιμετωπίζουν και άλλα κράτη-μέλη. Ιδιαίτερα σε σχέση με τις τελευταίε προκλήσει που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το κράτος δικαίου και την αποτελεσματική υλοποίηση του κράτους δικαίου και εφαρμογή του στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, εγώ τουλάχιστον διαρωτώ με μήπως θα έπρεπε να μετατρέψουμε το σημείο του ενδιαφέροντος των μελετών αυτών σε μια συγκριτική περισσότερο μελέτη των διαφορών χωρών. Εάν τηρούν δηλαδή την ε, αρχή του κράτους δικαίου. και στα περαιτέρω τμήματα της μελέτης βλέπουμε συμπεράσματα και συστάσεις σε δύο εκδοχές. Στη δεύτερη πιστεύω υπάρχει μια σύσταση ότι υπάρχει περιθώριο αναλογισμού για την προσεχή αντίστοιχη μελέτη. και επιπλέον αυτών των ερωτήσεων. Θέλω να ρωτήσω εάν έχουν εξετάσει αυτές οι αρχές την έκθεση για την καταπολέμηση διαφθοράς του 2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τη μόνη η οποία καταγράφει τις εξελίξεις μετά την απόφαση του 2011 για τις αιτήσεις εκθέσεις. Η Επιτροπή και ο Αντιπρόεδρος Τίμερμανς ξέρουμε ότι το 2015 απέστειλαν στον Πρόεδρο της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ επιστολή όπου δήλωνα ότι δεν πρόκειται να ακολουθήσουν αντίστοιχε εκθέσεις και ότι αντίθετα ε, τα ζητήματα της διαφθοράς και της καταπολέμησής της θα έμπαιναν στο, στις αιτήσεις εκθέσεις και στις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Βεβαίως, με βεβαίως ότι πρέπει να είναι ε, αδέκαστη και αντικειμενική η καταγραφή των εξελίξεων στις χώρες αυτές και τους, για τους μηχανισμούς τους, έτσι ώστε οι χώρες να είναι σε θέση και με βάση μια αντικειμενική αξιολόγηση να κρίνουν, να δουν ε, την πρόοδό τους, αλλά ταυτόχρονα να τη δουν και σε σχέση με άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις μου. Ευχαριστώ. <coughs> Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Η κυρία Μακοβέη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρώτη μου ερώτηση προς τους συντάκτες της ε, έρευνας, η πρώτη και μοναδική ερώτηση ουσιαστικά που έχουν απευθύνει είναι η εξή. Ε, πώς ε, καταλήξατε στα συμπεράσματα αυτά που μας παρουσιάσατε, παρακολουθήσατε αυτά που συνέβησαν το 2018 στις χώρες αυτές, αλλά και το 2017 και τα άλλα έτη είδατε το πόσο έχουν αλλάξει τα... πόσο έχει αλλάξει η λειτουργία του δικαστικού σώματος ε, σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με την κοινή των πολιτών. Είδατε τις ε, διαδηλώσεις, τις διαμαρτυρίες ε, των δικηγόρων, των εισαγγελέων που βγήκαν και διαμαρτυρήθηκαν. Γιατί αυτά τα οποία άκουσα στην έκθεση αυτά και παραθέτω ότι αναφέρεται ότι υπάρχει εγγύηση για την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος. Αυτά δεν ισχύουν. Μέχρι τέλη του 2016 ενδεχομένω να ισχύουν, αλλά από το 2016 και μετά έχουν ε, τροποποιηθεί σημαντικά τα πράγματα αυτά, προκειμένου ουσιαστικά η δικαιοσύνη να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της πολιτικής. Και γι' αυτό λοιπόν βγήκαν να διαδηλώσουν οι εισαγγελείς, οι δικαστές. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Η αλλαγή του ποινικού κώδικα και του κανονισμού λειτουργίας. Η διαφθορά. Προωθείται με τη μέθοδο αυτή. Και ουσιαστικά διευκολύνονται οι υποθέσεις διαφθοράς. Και γίνονται λοιπόν διάφορε διαδικασίε για την αλλαγή του ποινικού κώδικα. Είναι πιο εύκολε οι δωροδοκίε σήμερα πια. Και αυτά πλέον ε, δεν ε, καταχαρίζονται καν ως περίπτωση διαφθορά. Όταν κανείς δηλαδή στείλει τον αδερφό του, κάποιο μέρος της οικογένειάς του, για να κάνει μια δωροδοκία, δεν ισχύει αυτό πλέον, δεν θεωρείται αυτό καν πενικό αδίκημα. Ο πρόεδρος της ε, Ρουμανικής Γερουσίας θα πρέπει να έχει προσαχθεί εδώ και καιρό. Τι έγινε όμως όλο το 2017, έγινε μια τροπολογία προκειμένου να εξαιρεθεί η συγκεκριμένη ρήτρα από τον κώδικα. Αυτό τι σημαίνει ότι το ρουμανικό δίκαιο είτε πρόκειται για αστικό δίκαιο είτε πρόκειται για ποινικό δίκαιο διέπεται από ψεύδι. Μπορεί λοιπόν κανείς να λέει ό,τι θέλει, να λέει ψέματα και να μην μετράει ούτε καν ως πενικό αδίκημα. Ρωτώ λοιπόν, μιλήσατε με τον κόσμο, μιλήσατε με τον κόσμο που ξεχύθηκε στους δρόμους να διαδηλώσει το 2017 και το 2018, τον Ιανουάριο, τώρα πριν από λίγο, τώρα δα. Σας ε, προσκαλώ στην ε, τρίτο όροφο, θα δείτε μία έκθεση με φωτογραφίες των ανθρώπων αυτών που διαδηλώνουν και ο κόσμος λέει ότι θέλει δικαιοσύνη, δεν θέλει πλέον διαφθορά. Εγώ τα πράγματα τα βλέπω πολύ διαφορετικά από αυτά που μας προσφέρει η έρευνα αυτά. Είναι διαφορετική η εντύπωση μου και υπάρχουν πολλά παραδείγματα τα οποία μπορώ να σας δώσω σε ό,τι αφορά το ποινικό δίκαιο. Προτάσει ε, οι οποίες όταν ε, θα εγκριθούν τελικά θα κάνουν τη Ρουμανία παράδεισο εγκληματιών. Γιατί όπου γίνονται τέτοια πράγματα είναι πολύ απλή η παραβίαση του νόμου. Και φυσικά δεν υπάρχει συνέχεια. Υπάρχουν, για παράδειγμα, νόμοι, νόμοι οι οποίοι ορίζουν ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει η έρευνα χωρίς ε, ενημέρωση, πληροφόρηση του ατόμου κατά το οποίο γίνεται η έρευνα. Και έτσι λοιπόν συνεχίζεται η κατάσταση. Είναι πραγματικά αστείο. Αστεία αυτά που γίνονται τι αυτά που αλλάζουν και αυτό ασφαλώς θα επηρεάσει και τη δικαιοσύνη και τη συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό κρατών μελών. Όλα αυτά θα υπονομεύσουν ε, τις έρευνες, γιατί έρευνες που θα ξεκινήσουν, για παράδειγμα, στη Γερμανία ή στην Ισπανία, πολύ απλά θα παγώσουν στην ε, Ρουμανία. Για τον απλό λόγο, για παράδειγμα, ότι χρειάζεται ενημέρωση του κατηγορούμενου ο επικεφαλής των Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο επικεφαλής του κόμματος κατηγορείται για νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, κατάχρηση ευρωπαϊκών πόρων, πάνω από 120 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η έρευνα ξεκίνησε από τον Όλαφ, από την Όλαφ. Και φυσικά θέλουν να αλλάξουν τον κανονισμό σε εθνικό επίπεδο σε ό,τι αφορά την ε, Ρουμανία προκειμένου να την κλειτώσει και ο αρχηγός της αντιπολίτευσης. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν τη Ρουμανία, στη Ρουμανία το 2017-2018. Οι πολιτικοί δουλεύουν ο καθένας για την βάρτη του κατά των συμφερόντων της χώρας. Αλλά θέλουμε ισότητα ενώπιον του νόμου. Δεν μπορούμε να ανοιχτούμε κάποιοι να μην ε, προσάγονται λόγω της θέσης τους. Και μία μικρή ερώτηση θα θέλω να απευθύνω. Δεν σας γνωρίζω και δεν έχω ακούσει και την, το, την υπηρεσία σας, το ίδρυμά σας. Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω, έχετε ακούσει καθόλου την οδηγία για τα ίδια προϊόντα, για τα ίδια αγαθά. Πώς εφαρμόστηκε αυτή η οδηγία δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί και ουσιαστικά η οδηγία αυτή υφιστάται μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έξω σε γνωρίσω, κατά 99% δεν έχει εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο αυτή η οδηγία. Για την ε, την κατάσχεση ιδιωτικών ε, αγαθών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίση μίλησε και για θέματα δημοσίων προμηθειών σε ό,τι αφορά την διαφθορά και την ε, απάτη. Να σα υπενθυμίσω ότι πριν από κάποιε ημέρε ο κύριο ε, Τίμερμαν άσκησε για την υποχώρηση, για την επιδείνωση τη κατάσταση στη Ρουμανία σε ό,τι αφορά τα ποινικά δεδήματα, σε ό,τι αφορά την εξαρτησία του δικαστικού σώματο, σα παρακαλώ λοιπόν, Σα καλώ πραγματικά να βγείτε να μιλήσετε με τον κόσμο στου δρόμου. Καθημερινά βγαίνει ο κόσμο στον δρόμο. Ρωτήστε του ποια είναι η άποψή του. Και προ του συναδέλφου από την μόνιμη αντιπροσωπεία τη Βουλγαρία θα ήθελα να απευθύνω μια ερώτηση. Τα αποτελέσματα, τα απορίσματα καταχωρήσονται σε ένα track record. Με ερευνητικά στοιχεία. Δεν αναφέρονται λέξεις, αναφέρονται αριθμοί. Έχω ρωτήσω λοιπόν το εξή. Πόσα άτομα προσάχθησαν για υποθέσεις διαφθορά σε υψηλό επίπεδο στη χώρα σας και πόσοι μπήκαν στη φυλακή τελικά. Μάλιστα, η Πρόεδρος, θα ήθελα να δώσω το λόγο στους δύο συντάκτες της ε, έρευνας για να απαντήσουν. Ο κύριος Κρόιτς και ο αδελφό σα παρακαλώ να έχει πάρει το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ. Να απαντήσω σε αυτά που είπε η βουλευτή από την Βουλγαρία. Ο βουλευτή από την Βουλγαρία, συγγνώμη. Ενδεχομένω αυτό να μην προέκυψε επαρκώ από τι διαφάνειε, αλλά θα ήθελα να σα πω ότι στην έρευνά μα πιστεύουμε ότι υπάρχει τρόπος μιας πιο συγκριτικής ε, μεθόδου προσέγγισης για να καλύψουμε όλα τα κράτη-μέλη και υποδείξαμε κάποιες δυνατότητες. Ε, αναφέραμε το πακέτο της Ένωσης για τα πρωτοσδικαίωτα και τα δικαιώματα και επίσης σημειώνουμε ότι ναι, με αυτό δεν περιλαμβάνεται στη διαφάνεια, περιλαμβάνεται όμω την έκθεση. Αυτή η έκθεση για την καταπολέμηση τη διαφθορά όντω ε, διακόπη και νομίζω ότι θα έπρεπε να επανεισαχθεί προκειμένου ο μηχανισμός CVM να είναι πιο αποτελεσματικός σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση της κατάστασης σε όλα τα κρατημέλη. Επί του παράντος όμως πιστεύουμε ότι σημαντικό θα ήταν να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων σύμφωνα με τις πρόσφατες ε, συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν από ένα χρόνο. Αυτό θα πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο της τρέχουσας ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αν ε, διαπιστωθούν απτά αποτελέσματα για όλες αυτές τις συστάσεις, ενδεχομένως ε, θα μπορούσε να αντικατασταθεί ο τρέχον μηχανισμός με ένα διαφορετικό μηχανισμό, ένα διαφορετικό σύστημα το οποίο θα κάλυπτε όλα τα κράτη-μέλη. Και εγώ επιτρέψτε μου να προσθέσω τρεις κουβέντες για τα ερωτήματα που ακούσαμε σε ό,τι αφορά τη Βουλγαρία. Τη Ρουμανία, συγγνώμη. Είμαστε φυσικά ενήμεροι για τις διαδηλώσεις. Δεν ήμασταν εκεί φυσικά εκείνη την εποχή, αλλά ξέρουμε ότι έλαβαν προσφάτως χώρα διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες. Ε, το θέμα είναι πολύ ακαθόδες. Προκαλεί διχασμούς ε, το διαπιστώσαμε αυτό από τι συνομιλίε μα με διάφορα άτομα στη χώρα. Προσπαθούμε να αξιολογήσουμε τι συνέβη τα τελευταία 10 χρόνια. Και βάσει των αλλαγών που έγιναν την περίοδο αυτή, είχαμε την εντύπωση ότι υπάρχει περιθώριο πραγματικά για αισιοδοξία. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι δεν υπάρχει κίνδυνο επαναχώρηση και ξέρουμε ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και ελπίζω αυτό να προκύπτει από την εκθέσή μας. Στο σημείο αυτό θα περιοριστώ. Και αν έχετε περαιτέρω ερωτήσει, με χαρά μου να τι απαντήσω. Σα ευχαριστώ, λέει κυρία Μακοβέ. Δεν κατάλαβα τίποτα. ήρθαν σε επαφή, λέει, με κάποιους αρμόδιους στη χώρα, αλλά τι γίνεται με τη δικαιοσύνη, τι γίνεται με τη διαφθορά. Λένε θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υπάρξει κάθαστη δικαιοσύνη. Και έχουν περάσει τώρα δέκα χρόνια που τα λέμε αυτά. Θα πρέπει να γίνει η διάκριση μεταξύ εκτελεστικών υπηρεσιών όπως η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς και από την άλλη μεριά της πολιτικής, της πολιτικής βούλησης για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Και κάθε έκθεση λέει ότι να έχουμε στη Ρουμανία καταδίκες ε, υπουργών σε κάθριξη Ε, στη φυλακή μπήκαν και πρόεδροι ποδοσφαιρικών σωματείων και ένα σωρά, αλλά στη Βουλγαρία ή σε άλλες χώρες να Ανατολής και Κεντρικής ε, Ευρώπης δεν γίνεται τίποτα. Γιατί, γιατί δεν έγινε έρευνα, γιατί δεν υπάρχει διαφθορά. Επομένως, πάντα πάντα οι εκθέσεις ε, οι εκθέσεις αυτές οι CVM λένε ότι στη Ρουμανία αρχές κάνουν τη δουλειά τους Γι' αυτό και έχει μειωθεί η διαφθορά. Τώρα όμω τα λέει αρκετά αυστηρά τα πράγματα. Και λέει ότι υπάρχει πολιτική βούληση για κάτω το έλεγχο τη διαφθορά για να ξεμπλέξουμε τη διαφθορά μια και έξω επιτέλου. Μέχρι το 2016 κανείς δεν τολμούσε να τροποποιήσει την ε, νομοθεσία. Μέχρι που καταργούσαν και αδικήματα. Καθίστε να δείτε τις εκθέσεις της τελευταίας δεκαετίας. Αυτό το οποίο έλειπε, το πρόβλημα ήταν ακριβώς αυτό στην απουσία πολιτικής βούλησης. Αν θέλουν, μπορούν όμως οι πολιτικοί να κάνουν αυτό που πρέπει. Στη Ρουμανία εδώ και ένα χρόνο οι πολιτικοί θέλουν τώρα να προβούν στις σχετικές ενέργειες και σε κατάσχεση περιουσιών των εγκληματιών. Πρόεδρος. Ναι, θέλω και εγώ να πω δύο λόγια. Αν δούμε τις εκθέσεις αυτές της δεκαετίες, διερωτώμεθα τι έχει επιτευχθεί τελικά. Ναι, κάτι έχει προχωρήσει, το δέχομαι. Αλλά θα ήθελα πιο συγκεκριμένα πώς προχώρησαν, να μας πείτε. Ο μηχανισμός ε, πιστεύω ότι μπόρεσε να ενισχύσει τις δυνάμεις της αλλαγής της ε, χώρες και της δύο χώρες ε, και έχουν μπορέσει ορισμένοι να βρουν πραγματική στήριξη στο μηχανισμό αυτό. Ε, το πιστεύω ακράδαντα, έχει προχωρήσει και η πιο επαγγελματική οργάνωση της δημόσιας διοίκησης. Αν γίνεται αντίληπτο ότι ευρωπαϊκά κονδύλια πρέπει να χρησιμοποιούνται με βάση τους κανόνες, τέλος θα πρέπει να ε, ανακτώνται, επομένω στηρούνται οι κανόνες. Ήταν ατυχές ωστόσο ότι έγινε ταυτόχρονη ε, επεξεργασία των καταστάσεων των δύο κρατών, γιατί είναι διαφορετικά από αυτά που έχω δει εγώ, δηλαδή πιστεύω ότι είναι διαφορετικά τα δύο κράτη. Με το ε, ίδιο βαθμό εστίασης, με τα ίδια γυαλιά, τα κοιτάμε τα ε, δύο κράτη και αυτό ήταν ένα λάθος και αυτό το λάθος δεν το υπέστη παραδείγματι η Κροατία με τον ίδιο μηχανισμό και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει οι συστάσεις του μηχανισμού να προχωρήσουν περισσότερο, να αλλάξουν και βεβαίως πρέπει να κοιτάξουμε προς ποια κατεύθυνση πρέπει να μεταραγεί αυτό ο μηχανισμός, όχι μόνο για τα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά και για τα δύο κράτη σας, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Πρέπει να μεταξελιχθεί αυτό ο μηχανισμός και για τη Βουλγαρία και για τη Ρουμανία, γιατί χρειαζόμαστε και εκεί καλύτερα αποτελέσματα. Ένα πρόβλημα συγκεκριμένο, το οποίο και εσεί στήξατε, ρητά, ο βαθμός ε, της ε, αναγνώρισης πολιτικής βούληση σε όλα αυτά. Τα είδαμε σε μια ακρόαση που είχαμε κάνει, πολύ καλή ακρόαση. Και πρέπει να πω ότι δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι έχουμε επιτύχει στα δύο κράτη και αν είναι διαρκές το αποτέλεσμα. Το να είναι άνευ επιστροφής το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. η μονιμότητα του αποτελέσματος. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να μας πείτε σε ποιο βαθμό είναι και πού αυτά τα αποτελέσματα μόνιμα και χωρίς επιστροφή, χωρίς πίσω γυρίσματα. Και μας το είχε πει άλλωστε και ο Γενικός Εγγελέας στις ε, συζητήσεις μας στην Ακρόαση. Θέλουμε λοιπόν συγκεκριμένα να δούμε τι έχουν επιτύχει τα κράτη και όπως είπα μου είναι τόσο αδιαφορό ποιο έχει την κυβέρνηση. Ύστερα από 10 χρόνια παρακολούθηση κατάσταση. διαπιστώνω ότι δεν είναι πολύ σημαντικό το ποιο κόμμα θα έχει την κυβέρνηση, γιατί κάθε κυβέρνηση έχει τα σημεία τα πιο δυνατά και τα λιγότερο. Ε, Επομένω, το αποτέλεσμα λίγο πολύ είναι το ίδιο. Ναι και έρθει λοιπόν το ζήτημα της ε, καταπολέμησης διαφθοράς. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Από αυτά που κάνουμε, τι μπορεί να γίνει καλύτερα για να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Θα σας ακούσω βεβαίως και μετά θα ακούσουμε και τη Γενική Γραμματεία της Επιτροπής. Και βέβαια και τους εκπροσώπους των ε, μόνιμων αντιπροσωπιών. Οπωσδήποτε, αν θέλουν το λόγο. Η κυρία Μακοβέη πρώτα όμως. Το μικρόφωνο είναι κλειστό. Μικρόφωνο σα. Όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα, βοήθησε πάρα πολύ ο μηχανισμός CDM. Δεν θα είχαμε αυτή την υπηρεσία πια. Θα είχε διαλυθεί αυτή η υπηρεσία και άλλες θετικές αλλαγές. Δόξα τω Θεώ, ευτυχώς που έγινε αυτός ο μηχανισμός. Θα πρέπει όλα αυτά να συνεχιστούν μισού ό,τι παγιωθούν όλες αυτές οι αλλαγές. Βοήθησε επομένω ο μηχανισμός ελέγχου. Και ακούσαμε εδώ, ακούσαμε τις αγγελίες. Έχουμε, έχουμε νούμερα. Μιλούμε για 30 υπουργού που πήγανε φυλακή. Και 90, 90 βουλευτές που επίσης καταδικάστηκαν. Και 88 δικαστές και εισαγγελείς. Έχουμε αποτελέσματα και μπορούμε να αποδείξουμε ότι οι θεσμοί λειτουργούν. Όλα αυτά ίσω θα γινόντουσαν έτσι κι αλλιώ, αλλά δεν θα έρθει οι αλλαγέ, οι κινήσεις αυτέ από το CVM. Τι να κάνουν οι πολιτικοί σε πολλέ περιπτώσεις ε, δεν δέχθηκαν ε, την άρση της ασυλίας τους, αλλά είχαμε αλλαγές, έστω μετά από 10 χρόνια. Και πριν από δύο μέρες, ο αντιπρόεδρος Τίμερμανς είδατε τι είπε. και εμείς εκπροσωπούμε το λαό της χώρας. Και τελικά ο λαός εκπροσωπεί τη χώρα και γι' αυτό και κατέβηκαν στο πεζοδρόμιο να απαιτήσουν το να επικρατήσει δικαιοσύνη και σας ε, επαναλαμβάνω, ναι, βοήθησε ο μηχανισμός. Θέλουμε να συνεχιστεί ο έλεγχος αυτός από τον CVM. ναι, να ψήχισμα με αυτά τα ίδια τα, κριτήρια και ό,τι ισχύει σήμερα είναι, είναι μια χαρά. Και περιμένω να ακούσω και τι θα πει και ο εκπρόσωπος της Βουλγαρίας. Να σας ε, πω για αυτό που αναφέρεται όσον αφορά το ανέκλητο αυτών των αλλαγών. για την επιτευθύσα πρόοδο. Σας παραπέμπω σε αυτούς τους εξαντλητικούς πίνακες της εκθεσής μας όσον αφορά τις αλλαγέ στην νομοθεσία και στις δύο χώρες τελευταία δεκαετία. Και τώρα όσον την ε, παγίωση των ανέκλειθων αλλαγών είπαμε στην ε, εισήγησή μας, στην παρουσιασή μας ότι μπορούμε τώρα να ε, αισιοδοξούμε ότι θα πιάσουν τόπο αυτές οι αλλαγές και σίγουρα για την Ρουμανία τέλος πάντων. Πάντως, είναι σημαντικά αυτά τα στοιχεία που έχουμε για το πόσες καταδίκες έγιναν στη χώρα. Αυτό αποδεικνύει ότι εφαρμόζεται ο νόμος με συνέχεια και συνέπεια. Υπάρχει βέβαια η διαφθορά ανεξαρτήτως του ποιος κυβερνά. Αλλά είναι σημαντικό να διαπιστώνει κανείς ότι η αλλαγή κυβερνήσεω δεν οδηγεί σε ανάσχεση αυτής της πρόοδου. Γιατί αυτή η πορεία, αυτή η διαδρομή συνεχίστηκε παρά τι αλλαγέ κυβερνήσεων. Άρα θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι οι αλλαγές είναι μόνιμες. Η Βουλγαρία δε, είπαμε ότι έχει κάποιο πρόβλημα όσον αφορά την διενέργεια των δικών που πολλές φορές επηρεάζεται από την πολιτική κλπ. Άρα αυτό θα πρέπει να διορθωθεί και να αποκτήσει μια εξαρτησία δικαιοσύνη. Εγώ με τη σειρά μου να σας πω κάτι γενικότερο για το τι θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί για το αν είναι μόνιμες αυτές οι αλλαγές και για τις δύο χώρες. Και μάλλον το πιο σημαντικό στοιχείο εδώ είναι ότι οι προσδοκίες του κόσμου έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Είπαμε για τις ε, διαδηλώσεις, για, για, για τις διεκδικήσεις, για την, ε, την αγανάκτηση σε σχέση με τα πισωγυρίσματα. Πολύ σημαντικά αυτά όλα. Και ο μηχανισμός αυτός συνεργασίας και ελέγχου έχει στηρίξει αυτές τις ε, προσδοκίες όσον αφορά το τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, τι πρέπει να προβλέπει το δίκαιο, ε, συνειδητοποίηση. Όλα αυτά χωρίς τον μηχανισμό θα ήταν δύσκολο να κινηθούν. Βέβαια δεν είναι όλα τέλεια και ένας κίνδυνος ίσως είναι η διάψευση του κόσμου από τους ε, κυβερνώντες τους ή από άλλους πρόεδρους. Να θέλω να δώσω το λόγο και στους εκπροσώπους των κυβερνήσεων της βουλγαρικής κυβέρνησης καταρχάς. Παρακαλώ. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ως απάντηση στο ερώτημα για τις υποθέσεις διαφθοράς ε, δεν έχω μαζί μου στατιστικές, στατιστικά στοιχεία, αλλά μπορώ να σας πω ότι η ε, αριθμή των οριστικών καταδικών τα τελευταία τρία χρόνια είναι σταθερή. Αντίστοιχα και τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία έως το 2012, από το 2012 έως σήμερα έχουμε ένα ποσοστό καταδικών από 20 έως 72 για το οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά. Αλλά όπως είπα, λεπτομερή στοιχεία δεν έχω μαζί μου. Η πρόεδρος... Θα ήταν καλό αν έχετε συγκεκριμένα στοιχεία να μας τα στείλετε με μια επιστολή. Φαντάζομαι ότι θα έχετε κάτι, έτσι. Μπορείτε να μας το στείλετε. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πυρίνης και πάλι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να απαντήσω σε κάποια από τα σχόλια που κάνατε. Σε ό,τι αφορά το μονιμότητα των αλλαγών, θα ήθελα να αναφερθώ και εγώ σε αυτά που είπαν οι συντάκτε της ε, έρευνα σε ό,τι αφορά τι προσδοκίε. Αληθεύει όντω ότι η κοινωνία επιδεικνύει όχι μόνο προσδοκία πλέον, αλλά και αποφασιστικότητα απτή σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες ε, αλλαγές σε μια κατάσταση την οποία κρίνει συγκεκριτική. Και αυτό σε ό,τι αφορά τις τελευταίες ε, διαδηλώσεις μεγάλης έκτασης και στην πρωτεύουσα και στην υπόλοιπη χώρα σε ό,τι αφορά θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, ε, σε ό,τι αφορά θέματα οικοδόμησης ενός τερέτρου για σκι όπου όντως υπάρχουν σημαντικά στοιχεία που καταδεικνύουν ε, ότι υπάρχει θέματα, υπάρχουν θέματα διαφθοράς. Ε. Και ουσιαστικά αυτό που κατέστησε σαφές είναι ότι η εταιρεία που επενδύει είναι εταιρεία offshore που έχει δημιουργηθεί και συσταθεί με νόμιμο τρόπο. Άρα το αντεπιχείρημα είναι που είναι το πρόβλημα. Και σε αυτό αναφέρθηκα ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς θα πρέπει να θεωρηθεί και από πλευράς μηχανισμού. Μηχανισμού που επιτρέπει τις περιπτώσεις διαφοράς να ανακύψουν. πάντα θα πρέπει να κοιτάξουμε τις ε, συνθήκες τις οποίες ε, προέκυψε η, εκάθε, η εκάστοτε υπόθεση. Συμφωνώ με αυτούς που δημαρτύρονται και συμφωνώ ότι δεν μπορεί να έχει έδρα μια εταιρεία εκτός της χώρας, αλλά από νομικής άποψης αυτό δεν αποτελεί παραβίαση του νόσμου, άρα θα πρέπει να γίνουν αλλαγές και στις νομικές διαδικασίες και στις πρακτικές που επιτρέπονται για να αντιμετωπίσουμε αυτό που απασχολείται τώρα στην Επιτροπή μας, που είναι η κατάχρηση των ευρωπαϊκών πόρων ασφαλώς. Η κυρία Μάκοβα, αλλά τελευταία φορά και μετά κλείνει η συζήτηση, παρακαλώ. Νόμιζα ότι είχαμε παραπάνω χρόνο. Αλεθεύει αυτό που είπετε και... Συμφωνώ σε ένα στοιχείο σε ό,τι αφορά τη μελέτη. Αυτή το είπε και ο συνάδελφος. Τι είναι μόνιμο, τι είναι απαράλλακτο. Η επιθυμία του κόσμου να μην ε, εξαιρούμαστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις, η δικαιοσύνη να ευχεί για όλους με τον ίδιο τρόπο, για τους πολιτικούς και για τους κοινούς η χώρα μας να συνεχίσει να αναπτύσσεται. Να μην υπάρχει κατάχρηση ευρωπαϊκού χρήματος πλέον. Η Δάλος στη Συρία αποτελεί χώρα προέλευσης ό,τι αφορά τους μετανάστες. Ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους και διαδηλώνει. Μπορώ να σας δείξω εικόνες. Ανάβουν με τα κινητά τους ε, φως ε, και σχηματίζουν ε, την σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπετε εδώ πέρα στην εικόνα μια γυναίκα η οποία έχει τυλιχτεί στην Ευρωπαϊκή Σημαία και βλέπετε στο πρόσωπό της την απόγνωση και την απογοήτευση. Είναι σαφής η απογοήτευση λοιπόν στη Ρουμανία και είναι σαφές ότι λαμβάνουν χώρα σημαντικά πράγματα. Από τη Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, ποιος είναι παρόν να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και καταρχάς, καταρχάς, να καλωσορίσω το γεγονός ότι έγινε αυτή η έρευνα κατόπιν εντολής τη Επιτροπή σα, γιατί νομίζω ότι τα απορίσματα συνάδουν σε μεγάλο βαθμό και με την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπή προκειμένου να διαπιστώσουμε και να ελέγξουμε μετά από 10 χρόνια λειτουργία του μηχανισμού τι έχει πετύχει και τι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε. Θα θυμόσαστε ότι στι αρχέ του περσινού έτου, από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημοσιεύσαμε μια έκθεση η οποία ήταν διαφορετική στην προσέγγιση της σε σχέση με τις εκθέσεις του παρελθόντος. Έδωσε έτσι μια σύνοψη για τα 10 αυτά χρόνια, μια επισκόπηση για να δούμε ποιες ήταν πραγματικά οι αλλαγές. Επίσης, αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε μια κάπως διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με τη μελλοντική μας μεθοδολογία σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, μια περιορισμένη σειρά συστάσεων προκειμένου να ολοκληρωθεί και μηχανισμός CVM σε κάποια φάση εφόσον δεν υπήρχαν προφανώς βήματα προς τα πίσω, δεν υπήρχε επαναχώρηση σε ό,τι αφορά τα βασικά ορόσημα που είχαν τεθεί τα τελευταία χρόνια και τα οποία αξιολογήθηκαν τελευταία φορά πέρσι τον Ιανουάριο. Άρα θεωρώ ότι αυτή η επιθυμία να δούμε μακροπρόθεσμα τι επιτεύχθηκε το μηχανισμό είναι κοινή και από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σαφώς κάποια από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μηχανισμού σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τις ιδιαίτερες συνθήκες όταν συστάθηκε. Τότε αποτελούσε μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη μορφή συνεργασίας. Τώρα αυτό είναι λιγότερο συνήθιστο. Συνεργασία λοιπόν με τα κράτη-μέλη με πολύ εντελεχή τρόπο για θέματα πολύ ευαίσθητα για την κοινωνία. Ο τρόπος λοιπόν που επιτέλεσε τα καθήκοντα της Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξελισσόταν με την πάροδο του χρόνου. Και αυτό ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις να προκαλεί την αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μετακινηθεί υπερβολικά σε σχέση με τους αρχικούς στόχους, με τα αρχικά benchmarks. Εμείς θεωρούμε ωστόσο ότι έχουμε διατηρήσει τον πυρήνα των στόχων που είχαμε θέσει εξ αρχής. Κάποια από τα συγκεκριμένα στοιχεία τώρα τα οποία αναφέρατε. Θα θυμάστε, Πρόεδρε, ότι πέρσι το φθινόπωρο, όταν ο πρόεδρος Γιούγκερ έκανε την ε, ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, δήλωσε ότι φέτος το φθινόπωρο, το 2018 δηλαδή, θα υπέβαλε ένα έγγραφο σε σχέση με την εφαρμογή του κρατούς δικαίου. Και είμαι βέβαιος ότι στο σημείο αυτό η εμπειρία με το μηχανισμό CVM θα αποτελέσει πολύ σημαντική, σημαντικό παράγοντα Πιστεύω λοιπόν ότι η έκθεση και το πώς συνοψίζει τα αποτελέσματα του μηχανισμού CVM, τον αντίκτυπο του CVM, διαπιστώνει ότι ενδεχομένως να μην ήταν τέλειος, ενδεχομένως να μην έδωσε απάντηση σε όλα τα ερωτήματα. Το διαπιστώνουμε και εμείς αυτό. Ήταν άλλωστε πολύ απαιτητικά. Απαιτητικοί στόχοι που είχαν τεθεί. Φυσικά όλα αυτά εξαρτώνται ιδιαίτερως και από τη συνεργασία του πολιτικού κόσμου και των άλλων βασικών ε, παραγόντων της κοινωνίας. Θεωρούμε ότι βοηθήσαμε αυτούς τους παράγοντες να συνεργαστούν με τις ε, κυβερνήσεις, με την κοινωνία των πολιτών. Αυτό αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο στο μηχανισμό και στη λειτουργία το Τέλος, να πω ότι συμφωνούμε ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά το θέμα της μονιμότητας των αλλαγών και του track record. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε είναι πολύ δύσκολο να είμαστε βέβαιοι για όλα αυτά. Πάντα φυσικά θα υπάρχει ένα στοιχείο κριτικής για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα και το, την έκταση των αλλαγών. Αυτό εντοπίζεται προφανώς και με την ε, συνέχεια των track records των αλλαγών που έχουν επιτευχθεί. Αλλά προφανώς βλέπουμε και τις προσδοκίες και των μελών της Επιτροπής σας και των συντακτών της έκτασης Νομίζω ότι εξετάζοντας και τη δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαπιστώνουμε τη διάκριση γίνεται στους κόλπους των πολιτών μεταξύ των υποθέσεων αυτών και του αισθήματο του ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τουλάχιστον θεωρούμε ότι ο μηχανισμός EVM έδωσε κάποιες απαντήσεις και μας έκανε να διαπιστώσουμε πραγματικά αυτές τις αλλαγές. Ευχαριστώ. Θεωρούμε ότι ο μηχανισμός θα συνεχίσει λοιπόν. Αυτό που δεν συζητήσαμε ήταν το θέμα των ευρωπαϊκών πόρων. Κοιτώντα τα αριθμητικά στοιχεία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χαίρομαι που είναι εδώ και η κυρία Διαμού, η οποία είναι υπεύθυνη από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κοιτώντα λοιπόν τα αριθμητικά στοιχεία, βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι όλα εντάξει. Λες και υπάρχει διαφθορά παντού στις δύο χώρες, εκτός από τον, τους ευρωπαϊκούς πόρους. Εν πάση περιπτώσει, τα σημειώνουμε αυτά. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάρετε το λόγο για το, τη μεταξέλιξη ενδεχομένω του μηχανισμού. Προς το πού θα μπορούσε να κινηθεί ο μηχανισμός αυτός, τι πιστεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν θα θέλετε να τοποθετηθείτε, παρακαλώ. Um, intention Η πρόθεσή μας πέρσι με τη σχετική έκθεση ήταν το να τοποθετηθούμε με συγκεκριμένο τρόπο όσον αφορά αυτές τις συστάσεις. Οπότε και να έχουμε ορίσει ακριβώς το τι διαβήματα πρέπει να γίνουν, αλλά επίσης να απαιτήσουμε δέσμευση πολιτικής φύσεως. Άρα, ως αυτές τις να υπάρχει ακρίβεια. Πάντως, είχε απαιτηθεί προσπάθεια σημαντική. Και αυτό είναι τη στάση μας και Επίσης, με τις συστάσεις προσπαθούμε να κατευθύνουμε τη χώρα προς ε, κάποιο είδου θεσμικά πλαίσια, δημιουργία θεσμικών πλαισίων, τόσο ώστε να υπάρχει αυτού του είδους μία αναστρέψιμη κατάσταση ε, και ταυτόχρονα να αναλάβουν οι ίδιοι τις ευθύνες τους. Και όλες αυτές οι μεταβολές να είναι βιώσιμες μακρόπνοα. Αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει, ότι οι εμπλεκόμενοι, τα θεσμικά όργανα μέσα στα κράτη-μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες, να λάβουν τα ενία, να δεσμευτούν. Και με αυτή την προσέγγιση να έχουμε πραγματική ανάληψη των ενεργειών, των, των, των ευθυνών από τις, ε, τους θεσμούς αυτούς στα κράτη-μέλη. Θα σας ευχαριστώ, λίγο. Πρόεδρος. Ευχαριστώ, βέβαια. Για το τι θα κάνουμε περαιτέρω, που είναι και ένα κύριο ερώτημα, δεν έχω κάποια συγκεκριμένη απάντηση. Θα συνεχίσουμε τις επαφές μας, τις συζητήσεις μας, να βρούμε την καταλληλότερη λύση και βέβαια και με καλύτερα στοιχεία για τη χρήση των ευρωπαϊκών κονδύλων. Ευχαριστώ πολύ τους τάκτες της έκθεσης, τους ε, εκπροσώπους των μόνιμων αντιπροσωπιών Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Ευχαριστώ θέμα που ήρθατε. Ολοκληρώνουμε το θέμα αυτό στην ημερήσια μας διάταξη και προχωρούμε στο σημείο 4, ειδική έκθεση 2-2018, αποτελεσματικότητα της διαχείρισης τραπεζικών κρίσεων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κύριος Κέβιν Κάρντιφ από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι εδώ. Μια σύντομη παρουσίαση, 10-15 λεπτά. Κύριε Κάρντιφ, πολύ σύντομα, για να μας παρουσιάσετε την έκθεση, την ειδική έκθεση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάρντιφ, ευχαριστώ πολύ, θα είμαι σύντομος. Χαίρομαι που μπορούμε να παρουσιάσουμε την έκθεσή μας για τα συστήματα διαχείρισης κρίσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πρόκειται για, την τρίτη, ε, για τον τρίτο δημοσιονομικό έλεγχο. Έχει να κάνει με την εποπτεία των ε, τραπεζών. Καταρχάς, με την ειδική έκθεση του 2016 καλύφθηκε το θέμα αυτό. Το σύστημα αντιμετώπιση των τραπεζών σε περιπτώσεις όπου ε, η κατάσταση γίνεται πιο κρίσιμη με την τρέχουσα και ο κίνδυνος της αποτυχίας SRB, έκθεση που παρουσιάσαμε πριν από δύο εβδομάδες. Για την τρέχουσα, την τρέχοντα λοιπόν δημοσιονομικό έλεγχο, εξετάζουμε την διαχείριση με την μορφή της διαχείρισης κρίσης από πλευράς Ευρωπαϊκής Κεντρικής ε, Τράπεζας, ένα σχέδιο ε, διάσωσης τραπεζών σε περίπτωση κρίσεως, ε, εντοπισμό έγκαιρο των, ε, της υποβάθμισης και των συνθήκων γενικά των τραπεζών εάν ε, πηγαίνουν προς τα χείρο και βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ορίσει ένα σημαντικό πλαίσιο διαχείρισης κρίσεων τραπεζών, έχει οργανωθεί η ίδια, έχει εξασφαλίσει τους πόρους για τη διαχείριση των κρίσεων αλλά και για την εποπτεία των ε, τραπεζών ε, σε κατάσταση κρίσεως κατά τρόπο ικανοποιητικό. Έχουμε όμως και κάποια ευρήματα, κάποιες συστάσεις να διατυπώσουμε. Πρώτον, η ΕΚΤ έχει μια καλή διαδικασία όπως είπα. Η υποβολή των εκθέσεων, η παρακολούθηση, η εποπτεία είναι ικανοποιητικές. Υπάρχουν εργαλεία, υπάρχει καθοδήγηση για τις τράπεζες. Υπάρχουν κάποια όμως ζητήματα τα οποία για να αντιμετωπιστούν προτείνουμε η ΕΚΤ να δώσει περαιτέρω στοιχεία σε σχέση με την τυποποίηση των σχεδίων ε, διάσωσης, ανάκαμψης. Το λειτουργικό πλαίσιο της ΕΚΤ έχει κάποια σχεδιαστικά ελαττώματα, ε, όπως άλλωστε και προβλήματα στην ε, υλοποίηση στην πράξη. Δεν είναι το σύνολο των οδηγιών που έχει η ΕΚΤ επαρκές. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτά τα ελλείμματα, τα κενά, για να είναι και σε θέση και να αντιληφθεί ποια είναι τα νομικά ζητήματα, ποιες είναι οι προτεραιότητες δηλαδή και πώς μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τα διάφορα σενάρια. Αν έχουμε μια τράπεζα που κινδυνεύει από πτώχευση, είναι πιθανό να πτωχεύσει, θέλουμε Ε, καλύτερη κατάρτιση του προσωπικού και εργαλεία στη θέση του για τη διάγνωση και τη μετώπιση. Παρά τι συστάσει από την τελευταία έκθεση, δεν προχώρησε στα απαραίτητα μέτρα που είχαμε προτείνει εμεί η ΕΚΤ. Δεν θα υψέλθω σε λεπτομέρειε γιατί δεν έχω αρκετό χρόνο. Αλλά θέλω να σα το επισημάνω. Κάποιε από τι πληροφορίε που είχαμε ζητήσει δεν ε, δόθηκαν εξαντλητικά. Και άρα από αυτό το δημοσιονομικό έλεγχο βλέπουμε ότι δεν είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε λειτουργική αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης κρίσεων της ΕΚΤ στην πράξη και είχαμε αρκετά θετικές απαντήσεις. Για το σύστημα τώρα που έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για να λειτουργήσει το σύστημα αυτό πρέπει να έχει καλή συνεργασία η ΕΚΤ. Βλέπουμε ότι το πλαίσιο όπως ισχύει δεν είναι επαρκές. Δεν έχει τακτική ενημέρωση δεν υπάρχει ε, καθημερινή ενημέρωση για το σχεδιασμό των ε, τραπεζών που βρίσκονται σε κρίση, ο μηχανισμός ε, και το, το Διοικητικό Συμβούλιο Διχείρισης Κρίσεων. Χρειάζεται βελτίωση στη συνεργασία λοιπόν με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ίσως χρειαστούν και κάποιες αλλαγές νομικού χαρακτήρα. Ξέρετε ότι προτείναμε, όπως είχε ζητήσει το Συμβούλιο Διχείρισης Κρίσεων, να είναι πιο αυτοματοποιημένη η ενημέρωση. Αυτό το έχουμε στήσει και εμείς λοιπόν με τις συστάσεις μας. Αυτά πρόεδρε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Πυρίνσκι τώρα, εκ μέρους της συγκεκριτρίας. Yes, uh, Madam Chair, thank you for... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς η Γέρα Σέντερ είχε κάποια υποχρέωση να ζητήσει συγγνώμη, δεν μπορούσε να έρθει, αλλά ζήτησε να προσθέσω εγώ τι δικέ τη παρατηρήσεις. Υπάρχει αυτή η αξιολόγηση και είναι θετική όσον αφορά την αποτίμηση από πλευράς του Ελληνικού Συνεδρίου για αυτόν τον ενιαίο μηχανισμό. και ότι πάνε καλά τα πράγματα παρά το ότι υπάρχουν κάποια κενά όσον αφορά αυτήν την ε, ε, διαδικασία ανάκαμψη, ή σχεδιασμού τη ανάκαμψη. Πάντως χρειάζονται ακόμα κάποιες βελτιώσεις και θα ήθελα να σας διατυπώσω κάποιες ε, επιφυλάξει που έχουν ξαναδιατυπωθεί πρώτα-πρώτα ότι είχε κάποιους περιορισμούς κατά τον οικονομικό έλεγχο το Ελληνικό Συνέδριο γιατί δεν εδόθησαν από την Κεντρική Τράπεζα όλες οι πληροφορίες. Υπήρχε επομένω λογοκρισία όσον αφορά τις πληροφορίες που είχε πρόσβαση και σε πολλές περιπτώσεις είχε πρόβλημα το Ελληνικό Συνέδριο. Δεν μπόρεσε να φτάσει στα πιο ε, χρήσιμα συμπεράσματα για το σχεδιασμό της ανάκαμψης και αυτό βέβαια είναι απαράδεκτο γιατί αυτό δεν αποτελεί αξιολόγηση αφού λείπουν τα στοιχεία. Γι' αυτό και το ελεγκτικό συνεδρίο είπε ότι το να μπορέσει να έρθει σε συντονισμό και συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και την Κεντρική Τράπεζα αλλά και άλλες αρχές είναι κάτι το οποίο έμεινε ανολοκλήρωτο. Και όσον αφορά το, ε, αυτόν τον ενιαίο μηχανισμό ότι καλύφθηκε σε αυτή την έκθεση για το τύπο ενίος μηχανισμός όσον αφορά τον SRB και την Κεντρική Τράπεζα. Και ξεκαθαρίστηκε το πώς θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στις σχετικές και τις πληροφορίες. Λέει εδώ πέρα η έκθεση ότι η εποπτεία του 2017 ως κόστος ανήλθε στα 490 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε άλλη πληρέστερη αξιολόγηση υπολογισμό για τις δέουσες δαπάνες. τουλάχιστον ένα χρόνο βρισκόντουσαν σε κατάσταση διαχείρισης κρίσεων και περισσότερες τράπεζες είχαν κακές ε, επιδόσεις και ο SSM ήταν ε, ο μηχανισμός που χρησιμοποιήθηκε ως ε, εργαλείο. Το θέμα είναι σήμερα οι τράπεζες πόσο έτοιμες είναι. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι πιο σταθερή κατάσταση από ό,τι παλαιότερα, περί το 2008 δηλαδή. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σα πω ότι θέλω να καλωσορίσω τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Κεντρική Τράπεζα από τη φορά στην Επιτροπή μας. Δεν ε, μπορώ να σας ε, καλωσορίσω με το όνομά σας, αλλά εν πάση περιπτώσει σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αλέξη Φομβόιτ, ε, εκπροσωπώ τον ενιαίο μηχανισμό επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζα. Θα ήθελα να κάνω μια σύντομη παρέμβαση για να πω ότι εκτιμούμε ιδιαίτερα το έργο του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου για την ενίσχυση της ε, αποτελεσματικότητας της ε, τραπεζικής εποπτείας ε, της ΕΚΤ σε ό,τι αφορά την έκθεση αυτή, η ΕΚΤ έχει αποδεχτεί έξι από τις οκτώ συστάσεις και Θεωρούμε ότι η έκθεση δίνει πραγματικά επικοδομητικές συστάσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας μας. Γίνονται ήδη διάφορες εργασίες για την εφαρμογή των συστάσεων, μεταξύ άλλων τη συνεργασία με το σώμα του ενιαίου μηχανισμού και σε ό,τι την σχετική αξιολόγηση. Δύο από τις συστάσεις, ωστόσο, δεν έγιναν αποδεκτές. Σε ό,τι αφορά την ε, διανομή πληροφοριών και άλλα ζητήματα. Θεωρούμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεργάζεται επαρκώς σε ό,τι αφορά το πλαίσιο αυτό. Να σας δώσω κάποιες λεπτομέρειες τώρα αν θέλετε σε ό,τι αφορά την έκταση της συνεργασίας μας αυτής. Νομίζω ότι αφαιρώνουμε και έχουμε αφιερέωση και χρόνο και προσωπικό και ενέργεια για τα έγγραφα αυτά. Πάνω από 5.000 έγγραφα σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μας και 38 συναντήσεις και τηλεδιασκέψεις έγιναν και με την ομάδα ΕΚΑ όπου και δώσαμε περαιτέρω πληροφορίες, απαντήσεις σε, σε ό,τι αφορά τις ερωτήσεις του ενίου μηχανισμού. Και έτσι έλαβαν πληροφορίες, ε, καθώς και πληροφορίες σε σχέση με κάποιες τράπεζες κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Ωστόσο, οι πληροφορίες σε σχέση με τις τράπεζες ήταν ανωνυμοποιημένες ε, για να μην μπορεί να εντοπιστεί η ταυτότητα της κάθε μία τράπεζας. Άρα συνολικά το εύρος των πληροφοριών που χορηγήσαμε επαρκούσαν για να είναι επαρκείς και αναλυτικές οι εκθέσεις της ΕΚΑ για τα θέματα που την απασχολούσαν. Συνεργασία, κρίσεις, εντοπισμός κρίσεων, σχεδιασμός ανάκαμψης κτλ. Κλείνοντας λοιπόν, να επαναλαμβώ ότι είμαστε ευγνώμονες από πλευράς της ΕΚΤ προς την ΕΚΑ για την έκθεση της και λαμβάνουμε υπόψη τις συστάσεις τους και ελπίζουμε να συνεχίσει η καλή και αγαστή συνεργασία με τους αδελφούς της ΕΚΑ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα πράγματα είναι καλύτερα από ό,τι περίμενα. Νομίζω ότι είμαστε στην απαρχή μια μακρά και επικοδομητική συνεργασία από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλει κανεί το λόγο. Όχι. Πολύ ωραία ολοκληρώσαμε και το θέμα λοιπόν αυτό. Την πρώτη φορά λοιπόν κάναμε τη συζήτηση. Αν στη συνέχεια η συγκεκριά θέλει να το συζητήσουμε αυτό πιο επισταμένως, μπορεί να το επισημάνει. Θέλουμε να δώσουμε άλλους στα μέλη της Επιτροπής την ευκαιρία να συζητήσουν τα ζητήματα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν έγινε μια σύντομη παρουσίασε. Αλλά στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής ε, εξέτασης ενδεχομένω να το ξανακοιτάξουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαιρόμαστε που ήρθατε σήμερα. Και να περάσουμε στην ειδική έκθεση 3 του 2018 του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου έλεγχο της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών. Ο κύριος Μάρτης, ε, ο κύριος Μάρτης είναι μάλλον ε, ο υπεύθυνο από το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο και η δική μα συγγήτρια κυρία Γιάννα Σέντερ. Κύριε Μάτε, έχετε το λόγο και πάλι. Ευχαριστώ. Θα σας παρουσιάσω τα βασικά απορίσματα του ελέγχου μας για το πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει θέματα μακροοικονομικών ανισορροπιών. Να επικεντρωθώ βασικά στι συστάσεις. Να σας δώσω και το ιστορικό υπόβαθρο εν συντομία για να σας εξηγήσω γιατί κάναμε τις προτάσεις αυτές. Καταρχάς, πιστεύουμε ότι η σύνδεση μεταξύ της ανάλυσης ε, των μακροοικονομικών ανισορροπιών και των συστάσεων αναχώρα θα πρέπει να ενισχυθεί. Ο αδανικός τρόπος να γίνει αυτό είναι ο εξής. Έχουμε τα IDRs, in debt reviews, ανάλυση των μακροοικονομικών ανισορροπιών και μετά αξιολογούμε το πόσο σοβαρέ είναι αυτέ οι ανισορροπίε. Και στη συνέχεια συζητάμε τι διάφορε δυνατότητε εφαρμογή διάφορων πολιτικών και γίνεται μια ποσοτικοποίηση για το κατά πόσο θα είχε αποτέλεσμα η κάθε λύση για την αντιμετώπιση τη εκάστοτε ανισορροπία. Και στη συνέχεια προβαίνουμε στι συστάσει αναχώρα. Αυτό που προτείνουμε λοιπόν δεν είναι κάτι το εντελώ καινούριο. Στην αρχή της μακροοικονομική διαδικασία. ακριβώς αυτό εξετάζουμε. Ανάλυση, IDR, αξιολόγηση τη σοβαρότητας της περίπτωσης, ε, συζητήσει πολιτικέ και κάποιες ευρείε συστάσει, αν και ασφαλώ οι συγκεκριμένε συστάσει, ακολουθούν στην πορεία. Αν υπήρχε ένα πρόβλημα σε αυτή την αρχική ιδέα ήταν η έλλειψη παραγόντων μακροοικονομικής ε, δημοσιονομικής πολιτικής. Γιατί ο δίκτυπος της δημοσιονομικής πολιτικής και της πολιτικής εσόδων σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση ενισορροπιών θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη και θα μπορούσε να αποτελέσει αυτό εργαλείο αντιμετώπισης των ανισορροπιών. Αυτό έλειπε λοιπόν ως στοιχείο στην αρχική σύλληψη του σχεδίου και μια και έθιξε το θέμα το δημοσιονομικό. Αυτό δεν αναφέρεται και στη συνέχεια, με μία μόνο εξαίρεση. Εξαίρεση της ε, πρόσφατης ανάλυσης των πλονασμάτων στη Γερμανία και στο τι ανισορροπίες προκαλεί σε άλλα κρατημέλη αυτό. Θεωρώ ότι αποτέλεσε ένα θετικό στοιχείο αυτό, αλλά το θέμα της δημοσιονομικής πολιτικής νομίζω ότι δεν θα πρέπει να περιοριστεί μόνο στα πλαίσια του συμφώνου Σταθερότητα και ανάπτυξη. Αυτό περιορίζεται σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο. Δεν κοιτάει στο σύνολό τη τη δημοσιονομική πολιτική και τι ανισορροπίε τη. Κοιτάει μόνο το θέμα τη αναγωνιστικότητα σε σχέση με τη δημοσιονομική πολιτική. Το μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Οι δημοσιονομικέ ε, λοιπόν πολιτικέ θεωρώ ότι θα πρέπει να αποτελούν το σημείο του MIP. Να δούμε λοιπόν πώς διαμορφώθηκαν οι αρχικές ε, εκθέσεις ε, χρέωσης. Καταρχάς, αξιολόγηση των ανισορροπιών, πώς προέκυψαν από τα IDRs. E Αυτό αναφέρθηκε και στην ανακοίνωση της Επιτροπής. Επίσης και οι δυνατότητες πολιτικής έχουν αφαιρεθεί από τα IDRs. E Σε τελική ανάλυση, αντί να υπάρχουν ξεχωριστά έγγραφα, το οποίο το είχε ως σκοπό ο κανονισμός, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι έκανε, ξεκίνησε να εισαγάγει μία επισκόπηση, μία σύνοψη των ανισορροπιών αναχώρα και αυτό προφανώς επηρέασε την προβολή των στοιχείων αυτών, την προβολή και της όλης της δικασίας ε, MIP και τη δυνατότητα να πιστεί στο κοινό τι είδου δράσεις ήταν απαραίτητες. Η Επιτροπή λοιπόν ακολούθησε την εξή διαδικασία. Όλες οι διαδικασίες που προκύπτουν από την Ευρώπη 2020 έπρεπε να εξεταστούν και να αξιολογηθεί η σχετικότητά τους ως προς την δημοσιονομική πολιτική. Σε ό,τι αφορά μάλλον τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αμα... Μεσοπρόθεσμα όμω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό δεν έχει επιρροές στις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αν για παράδειγμα υπάρχει ανισορροπία στους τρέχοντες λογαριασμούς αλλά παράλληλα υπάρχει μια μακροπρόθεσμη μεταρρύθμιση. Αυτή η μακροπρόθεσμη μεταρρύθμιση θα έχει αποτελέσματα. Αλλά τέτοιου είδου αντιρρυφωτικές μεταρρυθμίσει. δύσκολα θα επηρεάσουν διάφορα μακροπρόθεσμα προβλήματα σε ό,τι αφορά του τρέχοντε λογαριασμού, ε, προβλήματα σε ό,τι αφορά το επενδυτικό περιβάλλον, για να αποφευχθούν ενδεχομένω κρίσει. Άρα, οι ίδιε οι συστάσει ουσιαστικά απομακρύνθηκαν από την ανάλυση και αυτό δεν βοηθάει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απαντησή τη δήλωσε ότι οι συστάσει αναχώρα δεν θα πρέπει να αποτυπώνουν μόνο την τελευταία σε βάθο ε, επισκόπηση. Θα πρέπει να περιλαμβάνουν και άλλα έγγραφα τη Επιτροπή και προηγούμενε μελέτε. ναι, ενδεχομένως. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβει ο κόσμος ε, γιατί αντιτυπώνεται μια συγκεκριμένη σύσταση ανά χώρα, εξετάζοντας ε, μια σειρά πληθώρα εγγράφων. Αυτή η απομάκρυνση λοιπόν των συστάσεων από την ανάλυση επηρεάζει, θεωρώ, το βαθμό της εφαρμογή των ενισορροπίων αυτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε και μας υπέβαλε πιστικά έγγραφα που καταδεικνύουν ότι ο βαθμός ε, ε, εφαρμογής είναι ουσιαστικά πολύ χαμηλός. Η επόμενη σύσταση που έχουμε να κάνουμε είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενεργοποιήσει μια αποτελεσματική διαδικασία για τις μακροπρόθεσμες ε, ανισορροπίες. Πώς αντιμετωπίζει τις ανισορροπίες αυτές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως τώρα. Δεν έχει συστήσει ποτέ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τέτοιο βήμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Έχει την ε, διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών, αλλά δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία. Δεν έχει ενεργοποιηθεί ποτέ η διαδικασία καθεαυτή και αυτό προφανώς ε, έχει δευτεί και από την έκθεση των πέντε πρόεδρων, όπου αναφέρεται ότι το διορθωτικό σκέλος, η διαδικασία δηλαδή αντιμετώπιση των ανισορροπιών, θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική και να τίθεται σε εφαρμογή μόλις εντοπίζονται τέτοιες ανισορροπίες. Και πρόσφατα επισημάθηκε ότι η χρήση όλων των εργαλείων για τη διαδικασία μικρομηχανικών ανισορροπιών συμπεριλαμβανομένη του διορθωτικού σκέλου είναι προς το συμφέρον της Ευρωζώνης. Επόμενη σύσταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει και να δημοσιεύει σαφή κριτήρια και διαδικασίε για την καταξινόμηση των ανισορροπιών. Εδώ χρειάζεται λοιπόν πιο πολύ σαφήνεια. Γιατί δεν μπορεί κάθε χώρα να μπει σε μια κατηγορία, γίνοντας, κάνοντας διακρίσεις μεταξύ των χωρών που είναι στην διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών, αλλά δεν υπάρχει κάποια διαδικασία και άλλων χωρών οι οποίες ενδεχομένως να ξεκινήσουν διαδικασίες στα πλαίσια του μηχανισμού αυτού. Αναγνωρίζουμε τα αφεντικά βήματα που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τα μεγάλα πλεονάσματα, για παράδειγμα, όταν αντιμετωπίζεται τέτοια ζητήματα αυτή η ανάλυση λοιπόν για τη Γερμανία θεωρούμε ότι ήταν ε, η κατάλληλη ενδεχομένω να καθυστέρησε, αλλά ήταν ασφαλώ ένα βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η δημοσιονομική αυτή η πολιτική θα πρέπει να, γίνει, να αναλύεται και σε χώρε που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Για παράδειγμα, αρνητικό επενδυτικό περιβάλλον, γιατί ο συνδεσμό είναι πραγματικά πολύ μεγάλο. Καλούμε επίση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βελτιώσει την ε, επικοινωνία να εξηγεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα Εθνικά Κοινοβούλια γιατί έχουν καταταχθεί οι χώρε σε μια συγκεκριμένη κατηγορία, γιατί έχουν γίνει συγκεκριμένε συστάσει. Αυτό θα ήταν ένα σωστό βήμα. Και να υπάρχει πιο σαφή σύνδεσμο, όπω σα είπα, μεταξύ ανάλυση και συστάσεων, για να βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει και υποστήριξη τελικά από το κοινό στις χώρες Για να είναι σαφές ότι η τρέχουσα μέθοδο δεν είναι πλέον κατάλληλη. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε περίπου 15 συστάσει σε 6 περίπου κατηγορίε Να πω δύο λόγια για τι δύο συστάσει που δεν δέχτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τα σαφή κριτήρια κατηγοριοποίηση Είναι η μία σύσταση που δεν δέχτηκε και κατά δεύτερον η άλλη σύσταση. Προτείνουμε στο επόμενο τη επόμενη αναθεώρηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει πρόταση για την αλλαγή των νομικών κειμένων που κατηγοροποιούν τις χώρες με υπερβολικές ανισορροπίες. Ως τώρα λοιπόν το κείμενο τι λέει. Το κείμενο για τις υπερβολικές ανισορροπίες διευκρινίζει ότι αν υπάρχουν πολύ σοβαρές τέτοιες ανισορροπίες και υπερβολική θα πρέπει να θέσει εφαρμογή ένα μηχανισμό υπερβολικών ανισορροπιών αλλά αυτό δεν προβλέπει υποχρέωση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει συστάσεις, αλλά απλά εκφράζει πολιτική βούληση να ακολουθηθεί ένα συγκεκριμένο τρόπος δράσης. Και μια και είσαστε ένας από τους συνομοθέτες, φαντάζομαι σας ενδιαφέρει το θέμα αυτό. Είτε δέχεστε αυτή την ερμηνεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είτε όχι. ενδεχομένω να πρέπει να γίνουν ε, τροποποίησεις, τροπολογίες στο κείμενο για να υπάρχει πιο καλή αποτύπωση στο κείμενο του τι συμβαίνει στην πράξη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Είχαμε συμφωνήσει να γίνει μια σύντομη παρουσίαση, εν πάση περιπτώσει. Ο συνάδελφο Πυρίνσκι έχει το λόγο. Uh, thank you, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομο αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχουμε ξεκάθαρη άποψη για αυτή τη διαδικασία των μακροοικονομικών ανισορροπιών από πλευράς της, του αρχικού σχεδιασμού, της σύλληψης της διαδικασίας σε σχέση με τη σημερινή συγκυρία της ε, ευρωπαϊκής οικονομίας. Όπως γνωρίζετε, η διαδικασία αυτή εισήχθη το 2011 λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Τότε είχαμε μεγάλα ελλείμματα, είχαμε τη φούσκα των ακινήτων, κίνδυνος, κίνδυνος. Οπότε αυτή η διαδικασία προβλεπόταν για να μην έχουμε επανάληψη της κρίσης. Και όλοι γνωρίζουμε, Πρόεδρε, ότι όλα αυτά εντάχθηκαν στο ευρωπαϊκό εξάμεινο, κάτι το οποίο είναι υποσύνεχή αναδιαμόρφωση. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο και εμείς θα πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει το εξάμεινο διότι θα πρέπει να προβληθεί περισσότερο, θα πρέπει να είναι η διαδικασία ε, πιο στεγανή στην εφαρμογή της. και πολύ καλά τα ε, είπαν οι προελίσσαντες ότι εδώ έχουμε ένα πρόβλημα, ένα πρόβλημα ενοιολογικό δηλαδή το πώς θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε, πώς θα μπορέσουμε να ορίσουμε τι θα πει ανισορροπία και πώς θα συνάδει η γενική, η όλη μας πολιτική με το σύμφωνο σταθερότητας και έτσι να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ανισορροπίες που αποτελούν ε, ένα πρόβλημα, έναν κίνδυνο και για το κάθε κράτος μέλος και για όλη την Ένωση επομένω. Αυτό είναι η δουλειά που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενδιαφέρει να ακούσουμε την άποψή τη. Όπως είπε το Ελληνικό Συνέδριο, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί Πώ εφαρμόζεται, πώ εκτελείται αυτή η διαδικασία, ποιε είναι οι επιπτώσει, τι γίνεται σε σχέση με τι συγκεκριμένε συστάσει. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, συμπέρασμα διαπίστωση τέλο πάντων που προκύπτει από την έκθεση. Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ και νομίζω ότι αυτό αποτελεί και ένα καθήκον το οποίο αναθέτουμε στον συνομοθέτη και ο συναδέλφος ε, ε, θα πάρει το λόγο μιας και το είχαμε υποσχεθεί από προηγουμένως από τη συζήτηση για την Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Um, Σα ευχαριστώ πολύ. Όλη η μέρα θα, θα, θα ήθελα να ακούω πρόθυμα για τις δύο αυτές χώρες. Ε, αυτή η ειδική έκθεση έρχεται σε πάρα πολύ σημαντική στιγμή και άρα θα πρέπει και εμείς να δούμε πώς η διαδικασία αυτή θα γίνει πιο κατανοητή και στον κόσμο αλλά και στους πολιτικούς στα κράτη-μέλη γιατί δεν αφορά μόνο το πώς θα εξασφαλίσουμε το ότι τα εθνικά κοινοβούλια ε, και όλοι στα κράτη-μέλη θα αναδέχονται τις ε, συστάσεις αλλά και να είναι εφαρμόσιμες αυτές οι συστάσεις όπως έγινε και σε παλαιότερες εκθέσεις. Ανά κράτος μέλος, να βλέπουμε τι πρόοδος υπάρχει. Και υπάρχει διαδικασία μεταξύ δημιουργία ισορροπίας και ενός προβλήματος σε ένα κράτος μέλος, το οποίο μπορεί να διορθωθεί με εσωτερική πολιτική. Και από την άλλη μεριά έχουμε το πώς θα διορθωθεί μια ανισορροπία που αποτελεί συστημικό κίνδυνο για όλο το σύστημα. Άρα έχουμε εδώ δύο ενότητες ε, δεδομένων, περιστατικών, στοιχείων που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η δημιουργία και οι κανόνες και όπως είπε και το συνέδριο πρέπει να τον λάβει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να κάνει το παραπέρα βήμα. Δηλαδή, τι γίνεται ιδίω στα μεγάλα κράτη-μέλη με τις ανισορροπίες, τι γίνεται με αυτή την διαδικασία και ό,τι κάνουμε να συνάδει με το σύμφωνα σταθερότητας. Να ισχύει διαδικασία κατά τον ίδιο τρόπο για μεγάλα και μικρά κράτη-μέλη και στην εφαρμογή της. Τώρα μελέτησα την έκθεση. Δεν ξέρω τι συμπέρασμα εξάγει το ελληνικό συνέδριο, αλλά πάντως το μοντέλο που τώρα έχουμε και αυτό μετά μια δεκαετία που ξέρουμε τι έγινε το μοντέλο λοιπόν είναι ότι έχει σχεδιαστεί αυτή η διαδικασία για τις ανισορροπίες. Τώρα πέρασε η κρίση. Έχουμε ρυθμούς αναπτύξης για την Ευρωζώνη, όμως θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την απρόσκοπτη εφαρμογή αυτών των κανόνων. Και διαβάζοντας την έκθεση, δεν είμαι σίγουρος. Και άκουσα και τι ελέγχθη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ακούσουν τη γνώμη της. Άρα είναι πολύ σημαντικό να δούμε εάν το μοντέλο, η διαδικασία που έχουμε σήμερα αν υπαρκεί για την επίλυση του προβλήματος. Θα πρέπει συνεχώς να εξελίσσουμε, να τροποποιούμε τη διαδικασία. Άρα, να δούμε σε τι συμπεράσματα μπορούμε να καταλήξουμε, να πάρουμε στα σοβαρά αυτή την έκθεση και τα συμπεράσματά της. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ, για να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Την εισηγήτρια, τους ε, βουλευτές που σχολιάσαν την έκθεση. Και θέλω, ξεκινώντας να πω ότι η Επιτροπή καλωσορίζει την έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου. Όπως είπαμε αρκετές φορές στην Επιτροπή σας, θα ήθελα να σημειώσω ότι είμαστε ταγμένοι στην διαφάνεια, τη λογοδοσία και βέβαια κάθε ε, έλεγχο που θα μας βοηθήσει στις προσπάθειές μας για βελτίωση της νομοθεσίας, εφαρμογής της και βέβαια στην περίπτωση αυτή την αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Θα είδατε από τις απαντήσεις της Επιτροπής, που είναι ενσωματωμένες στην έκθεση φαντάζομαι, πως η Επιτροπή κάνει δεκτές περισσότερες από τις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου και δεσμεύεται να τις υλοποιήσει. Πολλές από τις συστάσεις εστιάζονται στην ενίσχυση και βελτίωση πτυχών των μακρο, της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών, που επίσης απασχολεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναφέρθηκε άλλωστε επανειλημμένως μέσα στην έκθεση το ίδιο το γεγονό αυτό, όπως και από την συγκεκριτρία. Ε, επιτρέψτε μου επίσης να επισημάνω γενικότερα όπως ακούστηκε και από τον Ευρωβουλευτή νωρίτερα, ότι η εποπτεία αυτή για την αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών έχει καλύψει ένα σημαντικό κενό στην οικονομική εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν προϋπήρχε. Δεν υπήρχε δηλαδή πριν από την ε, κρίση αυτή η κάλυψη. Αυτή η διαδικασία λοιπόν καλύπτει ευρύ φάσμα των νέων. Εισήχθη το 2011 στο επίκεντρο της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτή η διαδικασία αντιμετώπιση μακροοικονομικών ανισορροπιών έχει ε, εξασφαλίσει τη δυνατότητα για προσαρμογές αποτελεσματικές και μόνιμες της οικονομίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα ε, μπορεί να συγκρατήσει και το κοινωνικό κόστος αυτών. Η προσαρμογή λοιπόν και ο επαναπροσδιορισμός ε, της στόχευσης τα τελευταία χρόνια είναι εντυπωσιακό Θέλω ιδιαίτερα να το τονίσω αυτό. Είναι μια σημαντική προσπάθεια των κρατών μελών. Και μπορούμε να διαπιστώσουμε ε, ότι ήταν εντυπωσιακά τα αποτελέσματα. Ταυτόχρονα όμως ο μηχανισμός αυτός ε, μακροοικονομικής ε, αντιμετώπιση μακροοικονομικών ανισορροπιών ε, στοχεύει και στη μακροοικονομική σταθερότητα. Επομένω, τώρα είμαστε στο 7ο έτος αυτής της διαδικασίας, 7ο έτος υλοποίησης της διαδικασίας. Η ίδια διαδικασία είναι σχετικά καινούρια, πρέπει να πω ακόμη. Η εμπειρία από τα πρώτα χρόνια υλοποίησης τη ε, διαδικασία μα λέει ότι έχει βοηθήσει στην ε, ευαισθητοποίηση για τις προκλήσεις και την προετοιμασία με κατάλληλες πολιτικές ώστε να ανταποκρινόμαστε στις κρίσεις. Η εποπτεία επίσης συνδέεται και με πιο αυστηρή εφαρμογή των συστάσεων και πρέπει να πω ότι μπορεί να μην ήταν πάντα οι πολιτικές δράσεις επαρκείς για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις, αλλά παρακολουθούμε πάντα την εφαρμογή. Επίσης, η εφαρμογή της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών ε, προχώρησε και με ε, προσαρμογές αναλόγως της εξέλιξης, ε, διδασκόμενοι δηλαδή στην πορεία και εμείς και τα κράτη-μέλη. Και γενικά η διαδικασία είναι αποδεκτή ικανοποιητικά, σταθερή από το σχεδιασμό της, χάρη στο σχεδιασμό της και την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δεν αμφισβητούνται και επί τη ευκαιρία θα συνεχιστεί η βελτίωση της υλοποίησης ε, της διαδικασίας και όπως είπα έχουμε κάνει δεκτές από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής περισσότερες συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου εκ των οποίων πολλές έχουν να κάνουν με την ενίσχυση κάποιων πτυχών που ήδη ε, ενισχύει και βελτιώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως σε παραδείγμα τη σαφή διασύνδεση μεταξύ των ε, συστάσεων αναχώρα και των ανισορροπιών. Σε αυτό πιστεύω ότι έχουμε πραγματοποιήσει πρόοδο και είμαστε διατεθειμένοι να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο στο πεδίο αυτό με βάση τις συστάσεις πάντα. Επίσης δεχόμαστε την σύσταση σε σχέση με τις ε, συνέπειες της μακροοικονομικής ε, πολιτικής. Το λαμβάνουμε και αυτό περισσότερο υπόψη στις, τα τελευταία χρόνια και επίσης η διάσταση της Ευρωζώνης έχει μεγαλύτερη σημασία πλέον για τις ανισορροπίες, για την εξετάσταση των ανισορροπιών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και έχει αρχίσει η Επιτροπή μας να εξετάζει αυτή τη διάσταση στις τελευταίες έρευνες της. Επίσης, κάποιες συστάσεις έχουν να κάνουν με την εξασφάλιση μιας καλής ανάλυσης. Η υλοποίηση από την Επιτροπή της Διαδικασίας και επαναλαμβάνω εδώ τα λόγια του ελεγκτικού συνεδρίου, στηρίζεται από μια καλή ανάλυση, αυτό είναι ήδη ένα εύσημο, από την έκθεση. Ταυτόχρονα βέβαια θα πρέπει να συνεχιστούν οι βελτιώσεις όπου χρειάζονται, όπου είναι δυνατές και εν προκειμένου είμαστε ευγνώμονες προς το δικαστήριο, που μας προς το ελεκτικό συνέδριο που μας υποδεικνύει τρόπους βελτίωσης. Επίσης το ελεκτικό συνέδριο καλεί για ενίσχυση της επικοινωνίας και της ορατότητας ε, της διαδικασίας. Συμφωνούμε και εμείς ότι είναι απαραίτητη και η επικοινωνία και η μεγαλύτερη προβολή της διαδικασίας ώστε να υλοποιείται και καλύτερα. Τώρα επιτρέψτε μου να το ασταθώ στις δύο υποσυστάσεις, οποίες δεν έχουμε κάνει δεκτές. Πρώτον, σύσταση του Λεκτικού Συνεδρίου για την κωδικοποίηση των κριτηρίων ταξικο, ταξινόμησης των ε, ανισορροπιών και δεύτερον, ε, για, την κωδικοποίηση των κριτηρίων που δεν οδηγούν σε κίνηση τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματο και εδώ, υπερβολικών ανισορροπιών. Και εδώ επιτρέψτε μου ε, τρία σχόλια και αρκετό περισσότερο χρόνο, γιατί είναι σημαντικό για να καταλάβουμε όλη την εικόνα, του γενικότερη κατάσταση. Η διαδικασία λοιπόν έχει ένα ευρύτατο φάσμα, ε, γιατί οι μακροοικονομικέ ανισορροπίε είναι περίπλοκα φαινόμενα και μπορούν να εκδηλώνεται με πολύ διαφορετικούς τρόπους, άλλωστε το έχουμε δει και από την ε, τελευταία κρίση. Αναλόγως της ε, συγκυρίας των περιστάσεων που ισχυροβέ στην κάθε ξεχωριστή χώρα. Και έτσι χρειάζεται μια ευέλικτη ένα ευέλικτο πλαίσιο αξιολόγησης. Απλοί κανόνες δεν πιστεύουμε ότι μπορούν να δώσουν κατάλληλη απάντηση στο περίπλοκο αυτό χαρακτήρα, στο περίπλοκο αυτό φαινόμενο και πρέπει να είμαστε Επιφυλακτική και προσεκτική ε, Δεν είναι σωστό δηλαδή πάντα να κάνουμε παραλληλισμούς μεταξύ της διαδικασίας περιπολικών ανισονοποιών και του MGP, του Συμφώνου Σταθερότητας, γιατί η εποπτεία της διαδικασία ανισορροπιών χρειάζεται κάποιες προσαρμογές που δεν μπορούν να περιοριστούν σε αποφάσεις που στηρίζονται μόνο σε αριθμητικά στοιχεία όπως αυτά του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Αυτό το τονίζω διότι το έκαναν δεκτό και οι συνομοθέτες, όπως το Κοινοβούλιο βέβαια, μεταξύ αυτών, όταν ε, θεσπίστηκε ο μηχανισμός του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Επίσης, ε, για την κωδικοποίηση πάντα των κριτηρίων ταξινόμησης των ανισορροπιών. Πάλι θεωρούμε ότι δεν είναι σύμφωνο με το πνεύμα του κανονισμού. Αυτό που προτείνεται, διότι αν κοιτάξουμε τον κανονισμό, ο κανονισμό δεν κωδικοποιεί την έννοια των ανισορροπιών ή των υπερβολικών ανισορροπιών. Απαιτεί όμως να λαμβάνεται υπόψη ένας μακροσκελής κατάλογος στοιχείων που χρησιμεύουν στην αξιολόγηση κάποιων οικονομικών στοιχείων. Αυτό είναι το πνεύμα του κανονισμού. Και σε αυτό θέλω να επιμείνω. Η τρίτη παρατήρηση για τις συστάσεις που δεν κάνουμε δεκτές. Η κίνηση, η θέση σε κίνηση της διαδικασίας υπερβολικών ανισορροπιών, εκεί όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντοπίζει τις υπερβολικές ανισορροπίες. Θέλω εδώ να τονίσω ότι δεν είναι κάτι το αυτοματοποιημένο για μας. Δηλαδή πρόκειται για, έναν, για μια λύση που μπορεί να επιλέξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά εμά και δεν θέλω να περάσω σε μακροσκελή εξήγηση της συνθήκης του κανονισμού και της συνάφειας μεταξύ κανονισμού και συνθήκης, αλλά σας παραπέμπω σε εξήγηση που έχουμε δώσει στις απαντήσεις μας στο ε, Box 3, εκεί όπου εξηγούμε γιατί θεωρούμε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το δικαίωμα της πρωτοβουλίας και διατηρεί διακριτική ευχέρεια για θέση ή μη σε κίνηση της διαδικασίας 121 παράγραφος 4 της συνθήκης. Από την ε, σύλληψη στο σχεδιασμό της διαδικασίας δεν έχει τεθεί σε κίνηση διαδικασία υπερβολικών ε, ανισορροπιών. Και θέλω αυτό να τονίσω και για τις χώρες υπερβολικών ανισορροπιών, γιατί υπάρχουν και άλλοι τρόποι παρακολούθησης στενής, ε, εποπτεία. και αυτό ισχύει και όταν εξετάζουμε την υλοποίηση. Η διαδικασία λοιπόν μακροοικονομικών ανισορροπιών έχει ρόλο να διαδραματίσει, μπορεί δηλαδή να οδηγήσει σε αλλαγή νοοτροπία τη κυβερνήση. Είναι κάτι το σημαντικό το οποίο δεν χρειάζεται, δεν πρέπει να αγνοήσουμε στη συζήτησή μα, πρέπει να παρασιοποιήσουμε. Και επίση, κυρία Πρόεδρε, Θέλω να επισημάνω τις απόψεις των ίδιων των κρατών μελών που τελικά εφαρμόζουν τις συστάσεις. Και το ελεκτικό συνέδριο έκανε μια πολύ χρήσιμη μελέτη με την έκθεσή του. Μια μελέτη λοιπόν όπου φαίνεται πως τα κράτη-μέλη κύριοι παραλήπτες αυτών των συστάσεων εν αξιολογούν τη διαδικασία την υλοποίηση διαδικασία μακροοικονομικών ισορροπιών θετικά. Πολλά είναι εκείνα τα οποία θεωρούν ότι έχει συμβάλει στην ανάπτυξη πολιτικών επιλογών και συζητήσεων διαλόγου στις χώρες τους και ότι ήταν πολύ σημαντικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 74% εν όλο των κρατών θεωρούν ότι είναι άκρος ή πάντως πολύ αποτελεσματική. Εδώ ολοκληρώνω. Ευχαριστώ το δικαστήριο για την έκθεση, για τις συστάσεις και πάλι για την επικοδομητική ε, συνεργασία για την υλοποίηση της ε, διαδικασίας ε, μακροοικονομικών ανισορροπιών. Είχαμε πει ότι πρέπει να είμαστε στα 10 με 15 λεπτά για το θέμα αυτό. Τώρα μας πιέζει ο χρόνος βεβαίως, γιατί έχουμε και άλλα θέματα που έχουν πάρει και καθυστέρηση που θα πρέπει να τα αφήσουμε. Τώρα πάμε στην ειδική έκθεση του 2018. Όσκαρ Χέριξ και ο κύριος Βόν για μας. Παρακαλώ κύριε Χέριξ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρο. Αγαπητοί κύριοι βουλευτές, θα προσπαθήσω πραγματικά να είμαι σύντομο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το 2016 ίδρυσαν αυτή την ε, κοινή πρωτοβουλία Jaspers σκοπός ήταν η εκπροσώπηση στις ευρωπαϊκές ε, περιφέρειες και υποστήριξη των ευρωπαϊκών τέτοιων πρωτοβουλίων. Αυτό που ήταν σημαντικό από οικονομικής άποψης. Μεταξύ 2006 και 2016 το πρόγραμμα Γιάσπερς έκλεισε ε, βοήθεια για 700 τέτοια προγράμματα και από οικονομικής πλευράς ε, είναι σημαντική η συνολική υπόστηριξη του Γιάσπερς για μεγάλα τέτοια προγράμματα 78 δις ευρώ. Συμμετείχε η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή με 46 εκατομμύρια. έπιση ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υποστηρίξε το Γιάσπερς με πάνω από 10 δισεκατομμύρια στην περίοδο 2007 έως 2013 και 10 δις ε, την επόμενη περίοδο. Σε ό,τι αφορά τη θεσμική σύσταση και τον σχεδιασμό του προγράμματος Γιάσπερς, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι τα βασικά, α, βασικοί στόχοι της πρωτοβουλίας και οι βασικοί φορείς δεν ορίζονται σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τις συμβάσεις εργασίας οι οποίες κρατεύτηκαν στην ΕΤΕΠ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και γι' αυτό, λοιπόν, υπάρχουν κάποια ερωτηματικά σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία αυτή. Η υποστήριξη Jaspers δεν ήταν αρκετά στοχοθετημένη. Δεν υπήρχαν, δηλαδή, τομεί προτεραιότητα για τα κράτη-μέλη. Και υπήρχε μεγάλο κίνδυνο έλλειψης ε, αμεροληψία ουσιαστικά σε ό,τι αφορά την περίοδο 2014-2020. Έχουμε μία νέα μεθοδολογία, μία νέα μέθοδο ε, ελέγχου της ανεξαρτησίας και ένα πρόγραμμα παροχής αρρωγής στα πλαίσια του Jaspers για μεγαλύτερο έλεγχο στη φάση στρατηγικού σχεδιασμού και κυρίως ορίζονται και κριτήρια αλλά και φάσεις της πρωτοβουλίας. Σε ό,τι αφορά τώρα τις πραγματικές ε, επιπτώσεις αυτών των μεγάλων προγραμμάτων, αυτό που διαπιστώνουμε είναι το εξής. Το Jaspers ε, οδηγεί σε καλύτερη επιλογή των προγραμμάτων και σε πιο γρήγορη εφαρμογή των προγραμμάτων είχε αντίκτυπο και στην ποιότητα των προγραμμάτων, το πρόγραμμα Jaspers, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το προγραμματιζόμενο κόστος και δεν υπήρχε επιρροή του Jaspers στα αποτελέσματα και στον αντίκτυπο και την ε, περίοδο εφαρμογής των προγραμμάτων. Το Jaspers επίσης δεν είχε αντίκτυπο σε ό,τι αφορά την εξάντληση των ευρωπαϊκών μέσων, γιατί υπήρχαν καθυστερήσεις σχεδόν σε όλα τα προγράμματα τα οποία έλεγξαμε και σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο στις διακριτικές ικανότητες των κρατών μελών. Ούτε εδώ διαπιστώσαμε μεγαλύτερη ανεξαρτησία των κρατών μελών λόγω της εφαρμογής του τζάσπερ. Και άρα οι συστάσεις μας είναι οι εξή ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εστιάσει το Jaspers ε, στη φάση σχεδιασμού είτε πρόκειται στη φάση εκκίνησης είτε στη μετέπειτα φάση του προγράμματος. Γιατί εκεί πραγματικά υπάρχει μεγαλύτερο αντίκτυπο Και αυτό που είναι σημαντικό είναι ο ρόλος και η ένταση της διαδικασία Jasper σε ό,τι αφορά την προσαρμογή αυτής στις ανάγκες των κρατών μελών προκειμένου να υπάρχει ανεξαρτησία, να μειώνει η εξάρτηση από το πρόγραμμα Jasper σταδιακά. Και τέλο να μιλήσω για το θέμα της εποπτείας και της αξιολόγησης. Το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο διαπίστωσε διάφορα προβλήματα σε ό,τι αφορά τι δραστηριότητε του προγράμματος Jasper στο σχεδιασμό, στην παρακολούθηση και στην αξιολόγηση, στη φάση του σχεδιασμού. Ποια ήταν τα προβλήματα. Υπερβολικά αισιόδοξε προβλέψει, σε ό,τι αφορά τον αριθμό των νέων προγραμμάτων προς υποστήριξη. Και έτσι, λοιπόν, μεταξύ 2014 και 2016 είχαμε μία αντίστροφη τάση σε ό,τι αφορά τους υπαλλήλους, ο αριθμό των υπαλλήλων ε, που αυξήθηκε σημαντικά και τον αριθμό των προγραμμάτων που μειώθηκε σημαντικά. Σε ό,τι αφορά το monitoring, ε, την παρακολούθηση, εδώ πέρα υπήρχαν προβλήματα σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα και την ε, αποδοτικότητα του Jaspers. Δεν υπάρχουν ε, ε, αξιόπιστα αριθμητικά στοιχεία ούτε σε ό,τι αφορά την εφαρμογή, ούτε σε αφορά το κόστος του Τζάσπερς. αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μας υπέβαλε τα στοιχεία αυτά. Και δεν μπορέσαμε να αξιολογήσουμε λοιπόν κατά πόσον η συνδρομή της ΕΤΕΠ στο Jaspers αντισταθμίστηκε από τα πλανεκτήματα του προγράμματος, δηλαδή κατά πόσον υπήρχε μια αναλογία σε ό,τι αφορά τα αμυνεκτήματα και τα πλεονεκτήματα και καταλήγουμε λοιπόν στις συστάσεις ε, στις οποίες προβήκαμε σε ό,τι αφορά την εισαγωγή ενός ε, εκτενούς ε, συστήματος ελέγχου και επιτήρηση για την επίτευξη των στόχων του Jaspers και επίση θα πρέπει να υπάρχει βελτιστοποίηση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην τρόπο λειτουργία του Jaspers να υπάρχει σωστή και αξιόπιστη εποπτεία των αποτελεσμάτων του Τζάσπερ. Και κλείνοντα κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να διαπιστώσω ότι από τις 12 συστάσεις μας, 9 έγιναν δεκτές απόλυτα και 3 εν μέρη μόνο. Άρα θεωρώ ότι υπήρχε σε μεγάλο βαθμό υποστήριξη από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, εδώ. Αυτή οι τομή συνεργασία ξέρουμε ότι ανοίγουν με το που γίνονται πιο ενδιαφέροντο. Ο κύριο Βόν έχει το λόγο. Είναι πολύ σημαντικό το Jaspers. Λέει και επειδή έχει επικρατήσει τελικά ότι αρχίζει από J να αποτελεί πρόγραμμα σημαντικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί είχαμε και άλλα που αρχίζουν από Τζέι. Λοιπόν, βλέπουμε ότι επικρίνεται το Jaspers από το ελεγκτικό συνέδριο. Όσον αφορά τον έλεγχο, όσον αφορά την αποδοτικότητα και ε, προκύπτει ότι θα πρέπει να γίνει βαθμία κατάργηση. Βέβαια έχει και κάποια θετικά η έκθεση. ότι είχε θετικές επιπτώσεις σε σχέση με τα έργα που πέρασαν από τον οικονομικό έλεγχο. Και επίσης είχαμε θετικές επιπτώσεις στα κράτη που εφαρμόστηκε το Jaspers. Αλλά είπαμε ότι έχει και άλλες αρνητικές ε, σκέψεις αυτή η έκθεση, οπότε θα πρέπει να απευθύνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μήπως θα μπορούσε να ε, σχολιάσει κάποιες από τις συστάσεις. Μας πει αν συμφωνεί, αν έχει κάποιες επιφυλάξεις, γιατί εγώ όταν μελέτησα αυτές τις συστάσεις διαπίστωσα ότι όταν δίνεται η υποστήριξη του Τζάσπερ σε κάποιο κράτος μέλος ότι ε, θα έπρεπε λέει, το ελληνικό συνέδριο να σταματάει εκεί το Τζάσπερς και τα κράτη-μέλη μόνα τους να αναλαμβάνουν τη συνέχιση των έργων. Και δεν ξέρω μήπως θα μπορούσε να υπάρχει υποκατάσταση του Τζάσπερς, ας πούμε να υπάρχει κάποιος τεχνική αρρώγη που να έχει καινούργια πρικοδότηση. Δεν ξέρω, εκτό αν η Επιτροπή συμφωνεί όσον αφορά τη βαθμία κατάργηση του Τζάσπερ και τι θα πρέπει να γίνει τότε να μα πούν. Ευχαριστώ, Γενική Διεύθυνση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ για το Ελληνικό συνέδριο και πρώτα πρώτα γενικόλογα για τον έλεγχο. Θετικά θεωρούμε τα όσα λέει η έκθεση και κατά την συνεργασία μας όλα πήγανε καλά με το συνέδριο. Για να δούμε λίγο το πλαίσιο αυτής της ιστορίας. Και όταν μιλούμε για βαθμία κατάργηση, ας σκεφτούμε και την ε, σταδιακή εφαρμογή του πριν από 10 χρόνια. Επρόκειτο για κάτι το οποίο δεν είχε προηγούμενο τα κράτη-μέλη 2004-2007 μπήκαν σε αυτή την υπόθεση και ε, λαμβάνουν πολλούς κοινοτικούς πόρους και άλλοι στην πρωταξιακή περίοδο. Και όλα αυτά για να εξασφαλιστεί η ποιότητα των έργων. Όποτε δεν υπήρχε η ιδέουσα διοικητική ικανότητα από τα κράτη-μέλη. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντοτε επιφυλάσσεται για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των έργων. Στη συνέχεια είχαμε πάνω από 500 έργα τα οποία αξιολογήθηκαν και υποστηρίχθηκαν και μιλούμε για 75 δις ευρώ σε πάρα πολύ σημαντικούς ε, τομείς. Και ε, βέβαια είχαμε δημιουργία δυνατοτήτων από τη, τον κρατικό μηχανισμό. Και έχουμε τώρα άλλα 600 έργα που προβλέπεται να δεχθούν την υποστήριξη. Τώρα, για την ε, αξιόλογηση του Jaspers. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία μηχανισμών υποστήριξης. Και συνεργαζόμαστε με την Τράπεζα Επενδύσεων, οπότε έτσι και ξεκινήσαμε την υπόθεση αυτή, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την εμπειρογνωμοσύνη της Τράπεζας Επενδύσεων για αυτά τα έργα. Επίσης δεν είναι θέμα μόνο της ε, DG, περιφερειακής πολιτικής, αλλά και άλλων. Move Connecting Europe, ε, προένταξε και άλλες υπηρεσίες της Κομισιόν, επομένως είναι συναρμόδιες. Τώρα, για το μόνο αφορά του συνεδρίου ακούσαμε και βέβαια συμφωνούμε ότι η ποιότητα των έργων ανέβηκε. Και έχουμε ένα δείγμα 20 έργων. Υπολογίζουμε τη συρρήγνωση της δαπάνης. Μιλούμε για 175 εκατομμύρια. Και αυτό το δείγμα αντιστοιχεί στο 3% των έργων που κάλυψε το Jaspers. Ήδη ακούσατε τι γίνεται όσον αφορά την συντόμευση του χρόνου έγκριση της Κομισιόν και αυτό είναι σημαντικό. Ε, το Jaspers τώρα από την στατιστικές μας βοηθά. Μας βοηθά να εγκρίνουμε κατά μέσο 85 μέρες. Και ένα από τα συμπεράσματα του ελληνικού συνεδρίου λέει ότι υπάρχουν και λιγότερα σφάλματα στα έργα που καλύπτει ο Jaspers. Από όλες τις συστάσεις ε, δεχόμαστε εν μέρη τρεις, ε, τις υπόλοιπες τις δεχόμαστε πλήρως, αλλά θα, ε, βεβαίως και θα πρέπει να υπάρξει αξιολόγηση, θα πρέπει να έχουμε καλύτερη εποπτεία, να υπάρχει επίσης καλύτερη στοχοθέτηση και έχουμε τώρα αυτά τα, αυτές τις ε, συστάσεις που δεχόμαστε μόνο εν μέρη πρώτα-πρώτα, τεχνικού χαρακτήρα σύσταση, αναφέρεται στο εξής θέμα. Πότε θα συντρέχει το Jaspers. Ε, βέβαια και συμφωνούμε ότι θα πρέπει από την αρχή, νωρίς. Αλλά όχι εάν έχουν συμφωνήσει για το έργο οι αρχές. γιατί άπαξ έχει γίνει η έγκριση και η συμφωνή η γνώμη των ε, τοπικών αρχών, τα πράγματα έχουν κρυθεί. Επίσης, όσον αφορά τις λεπτομέρειες λειτουργίας του Jaspers. Δεν θέλουμε να τις αναθεωρήσουμε επίσης. Πρόσβαση στα έγγραφα και όσον αφορά τις συμβατικές ρυθμίσεις με την Τράπεζα Επενδύσεων. Τώρα τι θα γίνει με τη βάση όλων αυτών. Όπως προαναφέρθηκε για αυτή την αμερόληπτη αξιολόγηση της ποιότητας Αυτό το έχουμε πει, το έχουμε συζητήσει με την Τράπεζα Επενδύσεων, οπότε ήδη αυτή η σύσταση έχει υλοποιηθεί, έχει εφαρμοστεί και κατά τα λοιπά η ΕΤΕ συντόμως θα υλοποιήσει τις ε, άλλες ε, συστάσεις. Και μέχρι να συνεδριάζει πάλι η Διευθύνουσα Επιτροπή, περιμένουμε να δούμε την υλοποίηση αυτών. Είπαμε για αυτή τη διαδρομή 10-12 ετών του Τζάσπερς, ποτέ δεν είναι πρόκειτο να αποτελέσει μόνιμο θεσμό. Αυτό είναι σημαντικό να μην το ξεχνάμε. Όχι, δεν μπορούμε τώρα να δεσμευτούμε για το πότε θα γίνει αυτή η βαθμία κατάργηση, αλλά πάντως μας βοηθά για την περίοδο 14-20 όσον αφορά την αξιολόγηση διαφόρων έργων και όχι μόνο για το συμβουλευτικό κομμάτι, αλλά και παραπέρα. και θα μπορούσαμε να φτάσουμε μέχρι το 2022. Ε, αυτό ας έχουμε κατά νου αυτή την περίοδο στρατηγική κατάρρησης. Πάντω συμφωνώ με αυτά τα οποία είπατε. Αυτά ε, λίγα λόγια για σχολιασμό αυτών των ε, επικρίσεων, των συστάσεων. Το Τζάσπες βοήθησε την ποιότητα των έργων στρατηγικού ενδιαφέροντος και συμφέροντος. Θα μπορούσαμε να κάτσουμε να αναλύσουμε βάσει συγκεκριμένων παραδειγμάτων έργων, αλλά τώρα έχει περάσει ώρα και δίγονται τέτοια πράγματα. Πρόεδρος. Ναι, ευχαριστώ. Είναι περασμένη όντω η ώρα. Μια σύντομη παρουσίαση θα πρέπει να είναι. Τέτοια ώρα. Σημείο εφευδομό. Ταξίδι στην Ελλάδα και αποστολή στην εβδομάδα την πράσινη της αποκριάς, της διακοπές. Θέλουμε να το προετοιμάσουμε. Έχουμε πίεση χρόνου γιατί κάποιοι από τους συμμετέχοντες εδώ που είναι πολύ σημαντικά στελέχη πρέπει να φύγουν κάποια στιγμή. Ας μου πούν λοιπόν όποιοι συνάδελφοι είναι εδώ που θέλουν τον λόγο. Είμαστε 7. Έχουμε πει ένα τόσο σημαντικό θέμα με τόσο σημαντικό κράτο, το οποίο πάει τόσο χρήμα. Καλό θα είναι να οργανώσουμε όσο δυνατόν καλύτερα την επίσκεψη. Διπλό ο στόχο. Τα 181 σχέδια προτεραιότητας του Ευρωτικού Ταμείου θέλουμε να δούμε πώ έχουν προχωρήσει. Πρόκειται για follow-up τη αποστολή του Σεπτεμβρίου του 2015 που είχαμε επισκεφθεί κάποια αυτά τα έργα και αυτή τη Αυτά τα έργα τα είχαμε συζητήσει με τις αρχές στην Αθήνα, μας είχαν, ε, συζητήσει για τις, μας είχαν μιλήσει για τις προεόδους, αλλά βέβαια τώρα θέλουμε να δούμε και τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη Λέσβο και το Ταμείο για τη Μετανάστευση. Θα επισκεφθούμε λοιπόν τη Λέσβο για μία μέρα. Έχουμε ο, να δούμε και θέματα Διευθυντικού Ταμείου αλλά και τον ε, προσφυγικό καταβλισμό στην Μόρια, hotspot και θέματα υποδοχής προσφύγων. Θα παρακαλέσω λοιπόν κύριε Μορτο να λάβετε στον λόγο και να μας ε, ενημερώσετε πολύ σύντομα και στο συγγνώμη για την πίεση χρόνου για τα θέματα στα οποία θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση. Παρακαλώ. Ε, πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Δύο λόγια, αν μου επιτρέπετε. Αν γυρίσουμε πίσω το ρολόι και δούμε ποια, είναι, ήταν η κατάσταση στην Ελλάδα ε, πριν από την μεταναστευτική κρίση και συγκρίνουμε με τα όσα γίνονται σήμερα, μπορούμε να πούμε ότι πολλά έχουν γίνει. Το 2015 η Ελλάδα δεν είχε ε, χώρους υποδοχής, δεν είχε εγκαταστάσεις ε, υποδοχής. Μέχρι το 2004 το πολύ ήταν πολύ κακές συνθήκες. Ακόμα και η αναγνώριση, η ταυτοποίηση των ε, προσφύγων και οι λοιπές διαδικασίες ήταν στα σπάργανα. Πολλά έχουν γίνει εντωμεταξύ και παρά ε, και πέραν και παρά την ε, δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Τουρκίας που άλλαξε άρδιν το σκηνικό με 95% λιγότερους, λιγότερες αφήξεις σχέση αυτά που είχαμε δει το 2015 βλέπουμε μια σημαντική προσπάθεια των αρχών της Ελλάδας κυρίως σε αυτό που θα ονόμαζα διαρθρωτικά μέτρα, διαρθρωτικές παρεμβάσεις για πιο καλά λειτουργούν σύστημα υποδοχής και ασύλου. Βλέπουμε κάποιες κέρδες εξελίξεις. Θα δείτε στη Λάσβο, παραδείγματι, Ε, λειτουργία hotspot σε συνεργασία κρατικών αρχών και υπηρεσιών κύριων φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτρέπει μια αποτελεσματική διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Έχουμε συστήματα δάκτυλοσκόπησης ε, που λειτουργούν στο 100% περίπου. Στην, ε, στην υπηρετική χώρα έχουμε ενίσχυση του δυναμικού υποδοχής 50.000 θέσεις. Στα νησιά Έχουμε επίσης ενίσχυση της υποστήριξης. Παραμένουν οι προκλήσεις. Αυτό οπωσδήποτε θα το παρατηρήσετε επανειλημμένο στη Μόρια. Πρόκειται για τον κατακλυσμό ο οποίο αντιμετωπίζει υπερπληθισμό αυτή τη στιγμή. Ένα από του λόγου είναι ότι και παρά την ε, δήλωση Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία δεν επιστρέφονται στην Τουρκία Σύριοι πρόσφυγε Σύριοι που έχουν έρθει στην Ελλάδα ε, παρά μόνο αυτοί οι οποίοι δέχονται να αποσύρουν την αίτηση ασύλου και να επαναπροωθηθούν στην Τουρκία. Λυπούμε που έχετε τόσο λίγο χρόνο. Αν τυχόν να σας περισσέψει έστω και μία ώρα, πηγαίνετε να δείτε το δημοτικό ε, τον δημοτικό καταβλισμό του Καράτεπε. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Η Μόρια έχει χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα της Ελλάδας. Το Καράτεπε το χρηματοδοτούμε εμείς μέσω του συστήματος έκτακτης βοήθειας σε συνεργασία απευθείας με την υπατιαρμοστία. Και τις τελευταίες μέρες, θα είναι ενδιαφέρον μάλιστα να το δείτε εσείς εκ πρώτης όψεως, από πρώτο χέρι, είδαμε αύξηση των αφήξεων στη Λέσβο και το συνολικό δυναμικό θεωρητικά είναι 5.000 θέσεις. Έχουμε φτάσει σε 7.000 αυτή τη στιγμή στο νησί. Και έτσι οι τοπικές αρχές αλλά και οι πολίτες του νησιού αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλη πίεση και πρέπει να πούμε ότι αυτό συμβαίνει ότι ταυτόχρονα σε μεγάλο βαθμό τα κονδύλια τα διαχειρίζεται η ε, κυβέρνηση της Ελλάδας σε κεντρικό επίπεδο, ύστερα από κάποιες δυσκολίες που ε, μας οδήγησε σε μια αργή εκκίνηση και το έχουμε ήδη συζητήσει, πρέπει να πω ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδο στους τελευταίους 12 μήνες από τις ελληνικές αρχές. Έχουν βελτιώσει τη δυνατότητα για απορρόφηση χρήση των κονδυλίων. Θα δείτε στη Μόρια πολλές προσπάθειες να προετοιμαστούν καλύτερα για να αντιμετωπίσουν τι δυσμενεί καιρικέ συνθήκες του χειμώνα. Ε, βεβαίως δεν έχουν καλυφθεί τα πάντα, αλλά πάντω είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από ένα χρόνο. Θα δείτε επίσης ε, προσπάθειε που στηρίζουμε και εμεί ε, με τη χρηματοδότησή μας να στηριχθούν οι πιο ευάλωτοι στη Μόργε. παραδείγματι. Υπάρχει μια ασφαλή ζώνη για τα μη συνοδευόμενα ανήλικα. Θα δείτε ότι προσφέρεται κατάλληλη στέγη για 70 μη συνοδευόμενους ασυνόδευτους ανηλίκους. Για τη συνολική χρηματοδότηση, μου επιτρέπετε δύο λόγια. Σημαντική χρηματοδότηση έχει διατεθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα μέχρι 600.000 ευρώ από τα προγράμματα ISF ε, και επίσης 600 εκατομμύρια, συγγνώμη, και 385 εκατομμύρια για κατεπίγουσα υποστήριξη, ε, χρηματοδότηση για ε, θέσεις ε, διαμονής, ξενοδοχεία και όλα αυτά τα οποία προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνθήκες του χειμώνα έχουν προβλεφθεί. είναι κάτι το οποίο είναι σκόπιμο να κοιτάξει κανεί, όπω άλλωστε έχουμε συστήσει να το κοιτάτε και όταν επισκέψετε την Τουρκία στι αντίστοιχε εγκαταστάσεις υποδοχής. Ε, υπηρεσίες επίσης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, διερμηνίας που δυστυχώς αυτή τη στιγμή έχουν πάψει γιατί δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση, πρόβλημα πρόσβαση στη χρηματοδότηση ε, για, το φορέα που, τις, ε, που διαχειρίζεται τις υπηρεσίες διερμηνίας και προσπαθεί να βρει μια λύση με τις εθνικές αρχές για την κατεπίγουσα υποστήριξη πέραν των δομών που έχουν εγκαθιδρύσει οι ευρωπαϊκές αρχές. Εμείς προσφέρουμε ε, συμπληρωματική υποστήριξη, πρόσωπο με πρόσωπο υποστήριξη, θα δείτε εκπροσώπου τη DG Home ε, εσωτερικών στη Λέσβο που είναι παρόν διαρκώ και θα σα εξηγήσει τι κάνει ακριβώ, τι προβλήματα αντιμετωπίζει, προσπαθώντα να στηρίξει και τι τοπικέ αρχέ, ακόμα και στο διάλογο που ενισχύεται χάρη στη βοήθειά του. Ε, πολλά μπορούν να γίνουν, επαναλαμβάνω, δεν ε, έχουμε φτάσει σε ένα τέλειο αποτέλεσμα, αλλά είναι πολύ σημαντική η βελτίωση και η πρόοδο στις τελευταίους 12 μήνες ε, από πλευρά των ελληνικών αρχών. Το πρόβλημα δεν είναι η χρηματοδότηση. Το κύριο πρόβλημα, κύρια δυσκολία, είναι όλη η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, η οποία είναι διαθέσιμη, να αξιοποιηθεί πλήρω και αποτελεσματικώς. Αυτή είναι η κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Ένα πράγμα που κάναμε και ολοκληρώσαμε το τέλος του 2017, ένα περίπλοκο αρκετά εγχείρημα καταγραφής των οικονομικών ε, στοιχείων, με ε, την προσπάθεια να καταγράψουμε και να απεικονίσουμε αποτελεσματικά και ε, με σαφήνεια την ε, χρήση των κονδυλίων, είτε απορροφώντα από εθνικέ αρχέ είτε από άλλου φορεί, δεν είναι εύκολο. Υπάρχει μια κοινότητα μη κυβερνητικών οργανώσεων που θα ήθελαν απευθεία να παίρνουν τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί το θεωρούν αυτό ευχερέστερο, χωρί όμω αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει μια μονιμότητα, μια σταθερότητα στι λύσει που μπορούμε να δώσουμε μακροπρόθεσμα, που επιδιώκουμε μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα να δώσουμε. Άρα πρέπει να έχουμε μια σταθερή χρηματοδότηση. Και επίση νομίζω ότι ο κεφαλή εκεί μπορεί να σα δώσει τις, ε, τα περισσότερα στοιχεία Έχω και άλλα βέβαια δεδομένα αν θέλετε να σας ενημερώσω για τις λεπτομέρειες της χρηματοδότησης. Τι χρηματοδοτούμε εμείς στο νησί. Βεβαίως, όπως είπα, είναι και ο εκπρόσωπός μας, ο συνάδελφος από την Digi Home και θα σας ενημερώσω λεπτομέρειες. Θα σας εύχομαι καλό ταξίδι και καλή επάνωδο. Ευχαριστώ. Βεβαίω, το fact sheet, ε, ο κατάλογο ε, που έχετε με τα στοιχεία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, Στι επισκέψεις και στην Τουρκία, το Λίβανο, την Ιορδανία μα έχουν απασχολήσει τα θέματα του Ταμείου για του πρόσφυγες, αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα που μα θα απασχολούν εν ώψη της επισκέψης στην Ελλάδα και βεβαίω και αυτά θα πρέπει να προετοιμάσουμε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ πάντω για την υποστήριξη σα. Πάντω, οι τρέχουσε εργασίε εντός εισαγωγικών είναι γεωργικά, διαρθρωτικό, ο ΠΚΠ θα επισκεφθούμε για το τομέα της γεωργίας. Καιρός είναι που δεν έχουμε πάει και από εκεί. Και περιμένουμε την ενημέρωση της κυρίας Χόχιμαν από την Γενική Διεύθυνση Γεωργίας. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και αγαπητοί κύριε Βουλευτές. Να πω ότι σας δώσαμε πληροφορία πληροφορίες γιατί ρωτήσατε πού βρισκόμαστε και πού είναι το ΠΚΠ σε ό,τι αφορά την, ε, ε, όλα αυτά τα τα στοιχεία αυτά. Κοιτάξαμε λοιπόν τα στοιχεία για το 2016 σε ό,τι αφορά την DG Agri. Όντω υπήρχε μεγάλο ποσοστό σφάλματος, 3,8%. Αλλά θα δείτε και στις πληροφορίες που σας δώσαμε ότι τρία από τα στα σημεία τα οποία περιλαμβάνονται είναι ότι ολοκληρώθηκαν δύο έλεγχοι και ένα έλεγχο είχε να κάνει με μια πρόορη ταξιοδότηση και αυτό ολοκληρώθηκε. Γιατί θεωρήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την Αμική Επιτροπή, ε, Υπηρεσία ότι δεν υπήρχε οποιοδήποτε σφάλμα στι πληρωμέ. Άρα, να σα πω ότι ναι, δεν υπήρχε υψηλό ποσοστό σφάλματο στι αιτήσει ε, δραστηριότητε ε, τρει από του πέντε ελέγχου έχουν ολοκληρωθεί, τρει από τι πέντε επιθεωρήσει. Και από ό,τι ξέρετε, όσο βρισκόμαστε σε διαδικασία αντίφαση ε, με το κράτο μέλος, αναμένουμε περαιτέρω πληροφορίε. Θα δείτε λοιπόν ότι στον πρώτο πυλώνα, στις άμεσες πληρωμέ, ε, υπάρχει βελτιωμένο σύστημα στην Ελλάδα, γιατί πραγματικά πριν από δύο χρόνια έγινε απόπειρα να βελτιωθεί το σύστημα και εξερεύθηκαν πάνω από 1,6 ε, εκατομμύρια άτομα που ατόμων που δικαιούταν περίθαλψη και να δούμε τι θα γίνει και το 2015. Και τελευταία είχαμε ένα θέμα με το ΠΚΠ που δεν είχε επαρκές ε, προσωπικός και έτσι λοιπόν δεν μπορούμε, ε, δεν είναι εύκολο να τηρείται ενήμερο το σύστημα. Ενδεχομένω λοιπόν αυτό δεν θέλουμε να το συζητήσουμε. Και τέλος είχαμε και κάποιες ε, αμφιβολίες σε ό,τι αφορά θέματα προώθησης στην αγορά και το άλλο από την οργανώση παραγωγών. Εδώ υπάρχει ένα σχεδίο δράσιο το οποίο είναι σε εξέλιξη για απορροκυπευτικά, για την πρόθεση αυτών, το οποίο σχετίζεται με ένα παλιό σύστημα πρόθεσης. Εξακολουθούν να υφίστανται λοιπόν ζητήματα, αλλά συνολικά μια πολύ βελτιωμένη κατάσταση για το ΠΚΠ από την προηγούμενη αποστολή. Ευχαριστώ. Η πρόεδρος. Υπάρχει λοιπόν αυτό το... Τι γίνεται μάλλον με το σχέδιο δράσης στην Ελλάδα. Το σχέδιο δράσης ολοκληρώθηκε και ενημερώθηκε το σύστημα ε, το, ε, για εξαιρέθηκαν 1,6 ε, δικαιούχοι, άρα θεωρούμε ότι ολοκληρώθηκε. Προκειμένου όμως το σύστημα να συνεχίσει να παραμείνει βιώσιμο, θα πρέπει να ενημερώνεται. Να ενημερώνεται κάθε τρία χρόνια τουλάχιστον. Τώρα έχουν περάσει δυόμιση χρόνια που έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο δράση. Ε, το θέμα λοιπόν είναι κατά πόσον θα υπάρξει επαρκές προσωπικό για να συνεχίσει την ενημέρωση του συστήματος. Κατά τα άλλα, θεωρούμε ότι το σχέδιο δράσεως ε, ολοκληρώθηκε και το ίδιο θεωρεί και το ελεκτικό συναντρίο για την έκθεση του 2015. Να ρωτήσω, λέει η Πρόεδρος, οι περικοπές στον τομέα του προσωπικού σε ό,τι αφορά τις ε, δράσεις ε, της ελληνικής κυβέρνησης, πώς απέδρασαν στο γεωργικό σύστημα και ε, χρειάστηκε κάποια προσπάθεια από το πλαίσιο αυτό. Είπατε 500.000 άτομα θα χρειάζονταν. Μπορείτε να μας δώσετε κάποια συγκεκριμένα ερευνητικά στοιχεία. <coughs> μιας και πρόκειται για κοινή διαχείριση, το προσωπικό της υπηρεσίας είναι αυτό που αποτελεί ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης, των ελληνικών αρχών καταρχάς. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι υπήρχε ανησυχία για την επαρκή στελέχνωση, για την ενημέρωση του συστήματος, όχι για το σχέδιο δράσης. Εκεί πέρα το προσωπικό ήταν επαρκές, αλλά εντωμεταξύ, όπως ξέρετε, όλα τα Όλες οι υπηρεσίες της ελληνικής κυβέρνησης έχουν πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη στεγλέχωση. Αυτό το παρακολουθούμε και το α, πρόγραμμα, το, το α, σύστημα διαπίστευσης. Στην Ελλάδα, λοιπόν, το Φεβρουάριο θα κοιτάξουμε τους συλλογισμό το 2017 και θα δούμε κατά πόσον το σώμα πιστοποίησης ε, πληρεί τα κριτήρια, μεταξύ των οποίων και η στελέχωση. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο στην παρούσα φάση. Προφανώς και αποτελεί αυτό ανησυχία, την οποία και συνεχίζουμε να παρακολουθούμε. Ευχαριστώ. Ερωτήσεις ε, που θα θέλετε να κάνουμε εκεί, που θα θέλετε να θέσουμε επί τόπου. Ε, as said, we have audit. Όπως σας είπα, βρίσκονται σε εξέλιξη διάφοροι έλεγχη και για παράδειγμα σε ό,τι αφορά το σύστημα LPIS. Ε, μια καλή ερώτηση θα ήταν αυτή που θέσατε μόλις σε εμάς. Ε, ποιος είναι ο αντίκτυπος ε, στο της στο προσωπικό. Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί και εμάς άλλωστε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό πρέπει να πω καταρχάς είναι ότι μου φαίνεται γελίο και λυπούμε αλλά μιλούμε για ψηφιακό μητρό. Έχω επισκεφθεί αρκετές φορές στην Ελλάδα και το 2015 βέβαια. Δεν νομίζω ότι είναι έτοιμο το ηλεκτρονικό μητρό. Η πρόεδρος... Ένα λεπτό. Είναι άλλο αυτό τώρα. Θα περιμένετε μετά, γιατί τώρα είμαστε στο κλιματολόγιο. Μετά θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Ίσως έχετε κάτι συγκεκριμένο για την εκπροσωπή. Ναι, αλλά για τα διαρθρωτικά ταμεία. Δεν φτάσαμε στα διαρθρωτικά. Δεν φτάσαμε. Στη Θεσσαλονίκη, λέει ο κ. Σιχώσκη, που επισκέφθηκα πριν από έξι μήνες, είδα πως ξεκίνησε η δουλειά, ακόμα δεν έχει τελειώσει, τίποτα δεν έχει προχωρήσει. Λίμνη χωρίς νερό είδαμε. Μας είπαν ότι θα ήταν σε ένα χρόνο. Ο δρόμος δεν έχει τελειώσει, η διάνοιξη ακόμα δεν έχει τελειώσει και για τους διερμηνείς επίσης έχουμε κάποιες πληροφορίες από εργαζομένους της Frontex και της EASO, που δεν είναι βέβαια υπάλληλοι, λέει ο μιλητής. Και μας λένε ότι για τη μετάφραση οι υπηρεσίες πληρώνουν το εξαπλάσιο πρέπει να εννοεί ο μιλητής από αυτό που κάνουμε εμείς όταν πληρώνουμε εμείς όταν έχουμε κάποιους στην Λέσβο για να μεταφράζουν. Δηλαδή πρέπει να χρησιμοποιεί κάποιες υπηρεσίες που προσφέρουν υπηρεσίες μετάφρασης για συγκεκριμένες γλώσσες η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά μου τα έχουν πει από το 2015, τίποτε δεν έχει αλλάξει. Είναι διάφορε συμβάσει οι οποίε είναι πολύ αμφιλεγόμενε. Η Πρόεδρος, καλά θα το ξανακοιτάξουμε αυτό, αλλά θα δώσω το λόγο στην κυρία Σλόιτερς και θα πω ότι έχουμε τα στοιχεία ο ε65, ο αυτοκινητόδρομος είναι το, στα έγγραφά μας, το ε, κτηματολόγιο, το μητρό, η λίμνη Κάρλα, περιβαλλοντικό ε, έργο, και βεβαίω θα μας ενημερώσετε για τις τελευταίες εξελίξεις και ό,τι άλλο έχει να κάνει με το Διευθυντικό Ταμείο και βέβαια με τη Λέσβο. Θα χρειαστεί κάπω να προσαρμοστεί το πρόγραμμα αναλόγω τη καταστάσεω, βεβαίως. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί βουλευτές, σας ευχαριστώ γιατί δείχνετε συνεχές ενδιαφέρον στην προσπάθειά μας που δεν είναι εύκολη. Όμως σιγά σιγά αποδίδει καρπούς. Και όπως προβλέπετε και σε άλλες εκθέσεις έχετε τώρα 10 έργα να συζητήσετε και να τα επισκεφθείτε. Είχαμε κατά 181, 2007-2013 ήταν το πλαίσιο το χρονικό της χρηματοδότησης που για χιλιάδες έργα και σας έχουν διαβάσει τα σχετικά έγγραφα όσον αφορά τα έργα που θα συζητήσετε. Εμείς γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι όσον αφορά το αποτέλεσμα βάζοντας υπόψη την ολοκλήρωσή τους και τη σχετική τεκμηρίωση, επίσης για τον ρυθμό ολοκλήρωσης, σχετική περίοδο για αυτό τα 181 έργα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τώρα έχουν ολοκληρωθεί όλα τα έργα. Υπάρχουν ορισμένα τα οποία εκκρεμούν, τα οποία συνεχίζονται. Είναι ανολοκλήρωτα. Ε, υπάρχει συγχρηματοδότηση από τις ελληνικές αρχές ή ε, λαμβάνουν χρηματοδότηση που ανήκει στην περίοδο 14-20 τώρα όσον αφορά τον αυτοκινητόδρομο τον ε65 μας ε, είπαν ότι το κεντρικό τμήμα του χρόνου άνοιξε στην κυκλοφορία άρα λειτουργεί και επισκεφθήκαμε το έργο στην Λιμνή Κάρλα το οποίο το συζητήσαμε τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και θα διαπιστώσετε ότι ολοκληρώθηκε το έργο όπως ακριβώς δεσμεύτηκαν οι αρχές ότι θα κάνουν στην προηγούμενη σας αποστολή. Τώρα σε σχέση με τις επισκέψεις που θα κάνετε για διάφορα έργα έχουμε ας πούμε την γραμμή τη θωρείας Λιανο Κλαδίου. Ολοκληρώθηκε με πόρους του Connecting Europe Facility. Και περί τα τέλη του 2018 θα παραδοθεί στην λειτουργία. Επίσης, η τρίτη γραμμή του μετρό των Αθηνών. Είναι πάρα πολύ μεγάλο έργο και τα τέλη του 2017 ολοκληρώθηκε η σχετική σύραγγα. Όμως, είχαμε ακόμα έργα που να γίνουν σε τρεις-τέσσερις σταθμούς. Εκεί και θα πάτε να δείτε τι γίνεται. Ε, μέχρι των οποίων και ο σταθμός του Πειραιά. Επίσης, όσον αφορά το κτηματολόγιο, και αυτό συνεχίζεται. Έχουμε πόρους από την περίοδο 2007-2013, αλλά θα υπάρξει συμπλήρωση από την περιοδο 2014 14-20. Εδώ βοήθησε το Jaspers και εμείς προβαίνουμε τώρα σε αξιολόγηση του τι γίνεται αυτά για μια συνοπτική εποπτεία του τι θα συζητήσετε, τι θα επισκεφθείτε και έχουμε τρεις συναδέλφους οι οποίοι έχουν αναλάβει τα σχετικά έργα. Και πάλι να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον σας στις προσπαθίες μας. Πρόεδρος. Εμείς σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη και η ερώτηση του κ. Στεχόφσκη είναι σίγουρα καλή και θα την ε, συμπεριλάβουμε. Θα μας ε, βοηθήσουν και οι βοηθοί να τι ε, λάβουμε υπόψη και να τι σημειώσουμε. Σα ευχαριστώ πολύ. Και για την ενημέρωση για την προπαρασκευαστική φάση. Είμαστε πέντε, ενδεχομένω να προσθεθούν και άλλοι δύο. Να σα παρακαλέσω όλου όσοι δηλώσατε ενδιαφέρον ε, να μην περιμένετε τελευταία στιγμή για να προετοιμαστείτε, γιατί έχουμε δουλειά. Ε, ολοκληρώσαμε λοιπόν το σημείο αυτό, να περάσουμε στο επόμενο σημείο, στο σημείο 8. Εδώ έχουμε έκθεση για την αποστολή στην Ουγγαρία. Έχετε την έκθεση μπροστά σας. Προσπαθήσαμε να την κάνουμε λίγο πιο εκτενή τη συζήτηση, γιατί είχε γίνει κάποια συζήτηση και προπαρασκευαστικά. Προσπαθήσαμε να ακούσουμε διάφορους, ε, διάφορες πτυχές για την ε, κατάσταση. Νομίζω ότι ήταν σημαντική η αποστολή και θετική διαπιστώσαμε ότι η Ουγγαρία αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα τα οποία θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και στο follow-up θα ήθελα λοιπόν στο σημείο αυτό να επιμείνω. Είχαμε μία συζήτηση και μία πιο συμβαστική συνάντηση με την Όλαφ για περιπτώσει απάτες. Αποστήλαμε διάφορα έγγραφα στη Βουδαπέστη. Πρόκειται για ένα περιβαλλοντικό έργο πρόγραμμα στην Βουδαπέστη και θέλουμε να συζητήσουμε και το θέμα των προμηθειών σε ό,τι αφορά το έργο αυτό, αλλά διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν και προβλήματα και σε άλλα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τις τέτοιες προμήθειες. Ε, διαπιστώσαμε ότι σε 36% των ε, περιπτώσεων, σε περίπτωση δημοσίων προμηθειών, ε, είναι ένας. Μία εταιρεία η οποία ωφέλεται από τους ευρωπαϊκούς πόρους. Να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας συνόδευσε στην όλη διαδικασία, κύριε Πέντα να σας δώσω το λόγο, κυρίως να μιλήσετε για το θέμα των ε, προμηθειών και θα πρέπει να κοιτάξουμε και το θέμα της επιλογής των προγραμμάτων, το οποίο δεν μας απασχόλησε έως τώρα, γιατί οι αρχές ήταν παρούσες μόνο για ένα τέτοιο project και τελικά δεν ξέρουμε πώς γίνεται η επιλογή, αλλά θέλουμε σε κάθε περίπτωση να διευκρινίσουμε το θέμα αυτό. Σας παρακαλώ λοιπόν γιατί αφωτίστε μας λίγο. Κύριε Μπέντε, να σας δώσουμε το λόγο και φυσικά αν οι συνάδελφοι θέλουν να κάνουν ερωτήσεις, ε, θα πάρουν το λόγο μετά. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί βουλευτές. Εισαγωγικά, να πω δύο λόγια για την ίδια την έκθεση και πώς την ε, ερμηνεύουμε εμεί το σύντομο χρονικό διάστημα που είχαμε στη διάθεσή μας. Είναι σαφής, νομίζω, η έκθεση σε ό,τι αφορά τις επισκέψεις που κάνατε. Νομίζω ότι τις αποτυπώνει σωστά και νομίζω ότι αποτυπώνει σωστά και τη δική μας ε, θεώρηση για τα προγράμματα δευτικών ταμείων στην Ουγγαρία. Καταρχάς, ε, σε ό,τι αφορά τη σημασία των διευθυντικών ταμείων, αναφέρεστε άλλωστε στο σημείο αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να επαναλάβουμε στο σημείο αυτό το πόσο σημαντικά είναι για την ευρωπαϊκή οικονομία τα ταμεία συνοχή και τα σωστικά ταμεία. Η ροή ήταν καλή στην περίοδο 2007-2013. Πάνω ε, του 100% των μέσων δαπανήθηκαν. Και η, ε, η Ουγγρική κυβέρνηση τώρα περιμένει μια επιστροφή της τάξης του 5%. Αυτά τα ονομάζετε επιτυχή και ολοκληρωμένα προγράμματα στην εκθέσή σας. Αυτό καταδεικνύει ότι ήταν καλή η απορρόφηση των πόρων και η δαπάνη στα προγράμματα. Ωστόσο, θα πρέπει να διευκρινίσουμε και άλλο ένα σημείο εδώ. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε το εξή. Παρά το γεγονό ότι τα ταμεία συνοχή και τα δερφωτικά ταμεία φτιάσαν το 3%, το 3 στην περίοδο 2007 έως 2013 και χωρίς ε, τα επενδυτικά αυτά τα ποσοστά θα είμαστε στο 13% διαπιστώνουμε ότι η σύγκληση η εξωτερική αλλά και εσωτερική δεν είναι αυτή η οποία ελπίζαμε και προσδοκούσαμε στο πλαίσιο των συζητήσεων για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο Ευρώπη 2020 αυτό που μας απασχολεί ιδιαίτερως είναι η Ουγγαρία σε σχέση με τις γειτονικέ ε, χώρες και τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και την Κροατία δεν πέτυχε το στόχο της πιο γρήγορης σύγκλησης. Αυτό τι σημαίνει ότι η ανάθεση των μέσων είναι, δεν είναι η βέλτιστη. Η έκθεσή σας και πάλι αποτυπώνει ακριβώς αυτό το πρόβλημα σε επίπεδο προγραμμάτων. Και τίθεται λοιπόν το ερώτημα της ποιότητας των δημοσίων δαπανών. Είναι άραγε ιδανική. Κάνετε και ερωτήσεις που αξίζει τον κόπο η δαπάνη των χρημάτων, value for money ή για παράδειγμα μονομενα προγράμματα για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής σύγκλησης. Όπως ξέρετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοιτά σε περιπτώσεις ε, κοινή διαχείρισης, ε, όχι τόσο πολύ σε πρώτη φάση τα προγράμματα, κοιτάμε τα προγράμματα, αλλά και εμεί ουσιαστικά παρόμοια ερωτήματα θέτουμε και ίδιες εμπορίες έχουμε. θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι σε σχέση με την περίοδο 2007-2013 έχουν γίνει και αλλαγές με βοήθεια του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου ασφαλώς. Πλέον δηλαδή έχουμε μια προγραμματική περίοδο η οποία επιμένει σε θέματα απλούστευσης και απλοποίησης και επικεντρώνεται στα αποτελέσματα. Ελπίζουμε αυτά να είναι θετικά στοιχεία και οι επενδύσεις οι οποίες ενδεχομένως να έχουν σημειώσει κάποιες ε, μείωση Μάλλον οι επενδύσεις που δεν έχουν μεγάλο αποτελέσματα και μεγάλη απόδοση έχουν μειωθεί. Ασφαλώς αυτό είναι κάτι που παίρνει χρόνο. Αλλά νομίζω ότι η εστίαση στα αποτελέσματα είναι η σωστή κατεύθυνση. Το τρίτο σημείο το οποίο ήθελα να θέσω και το θέξατε κι εσείς κυρία Πρόεδρε έχει να κάνει με τις δημόσιες προμήθειες. Σωστά το υπογραμμίσατε αυτό στην έκθεσή σας. και καταλήγεται ουσιαστικά στα ίδια αποτελέσματα όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ουσιαστικά το θέμα των δημοσίων συμβάσεων μας απασχολεί σε δύο επίπεδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά Τη συζήτησή μα με την, Ευρωπαϊκή, με την Ουγγρική κυβέρνηση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξημένου και την ποιότητα των δημοσίων συμβάσεων και το πώ διοργανώνονται η ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. Αυτό το αναφέρουμε σε κάθε έκθεση από την αρχή του εξαμήνου και επικρίνουμε κυρίως το πώς οι διαγωνισμοί γίνονται ουσιαστικά με έναν και μόνο με μία μόνο, μόνη εταιρεία ως υποψηφία. Πριν από μία, ένα μήνα έγινε μία επίσκεψη στην ε, Ουγγαρία και μισή μέρα αφιερώθηκε ιδιαίτερα στο θέμα των δημοσίων συμβάσεων. Για να γίνουν συγκεκριμένες ε, βελτιώσεις ε, σε ό,τι αφορά το θέμα των δημοσίων συμβάσεων. Και γιατί λέω στην πράξη, γιατί θεωρητικά εφαρμόζονται οι σχετικές νομοθεσίες. Και ουσιαστικά πλέον πρέπει να βελτιωθεί η υλοποίηση. Το δεύτερο επίπεδο που μας απασχολεί είναι το θέμα των ελέγχων και των επιθεωρήσεων. Και ο συνάδελφός μου ενδεχομένω ε, να θέλει να πάρει το λόγο για το θέμα αυτό. Αλλά μας απασχολούν ε, πολλά λάθη στο θέμα των δημοσίων συμβάσεων, πολλά σφάλματα και πολλές διορθώσεις ε, σε κάθε περίπτωση. Και αυτό εσείς αναφέρεστε στα αποθεματικά που προβλέπονται για τις, ε, τα προγράμματα αυτά. Πέντε από αυτά τα αποθεματικά προκύπτουν από προβλήματα ακριβώς σε θέματα δημοσίων συμβάσεων. Αυτό τι σημαίνει ότι προσπαθήσαμε να τα αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά με στενή συνεργασία με τις εγκρικές αρχές. Το τέταρτο θέμα που ήθελα να αναφέρω έχει να κάνει με το σύστημα ελέγχου και επιθεωρήσεων. Σωστά επισημαίνεται ότι στην Ουγγαρία είχαμε μεγάλο ποσοστό δημοσιονομικών διορθώσεων. Ένα δις στην περίοδο 2007-2013. Πιστεύουμε παρόλα αυτά ότι μπορούμε να πούμε ότι το συνολικό σύστημα ελέγχου και επιθεωρήσεων λειτουργεί αρκετά καλά, γιατί καταφέραμε να διαπιστώσουμε και το ποσοστό σφαλμάτων αυτό. Το μόνο αρνητικό είναι ότι όλα αυτά ήρθαν κάπως καθυστερημένα. Θα θέλαμε αυτές οι διορθώσεις από πλευράς των Ουγγρικών αρχών να είχαν γίνει πιο νωρίς και να μην χρειαστεί δηλαδή πρώτα να τα επισημάνει όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ο ΟΛΑΦ, το Ελεκτικό Συνέδριο. Τελευταίο σημείο το οποίο ήθελα να αναφέρω, αν μου επιτρέπετε, έχει να κάνει με ένα project. Να σας αναφέρω τι έγινε το μετρό υπαριθμών 4, γραμμή υπαριθμών 4 έγινε μια συζήτηση στη Βουδαπέστη και ρωτήσαμε γιατί καθίστερε τόσο πολύ το όλο πρόγραμμα και μήπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συμμετείχε όσο θα έπρεπε. Δυστυχώς, στη συγκεκριμένη περίπτωση εξακολουθούν να είναι σε εξέλιξη έρευνες. Οι Ουγγρικές Αρχές έχουν υποβάλει όλο το πρόγραμμα σε έρευνα και τα δικαστήρια ακόμα δεν έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες τους. Στην επόμενη λοιπόν ημερομηνία για διαπραγμάτευση είναι ο Σεπτέμβριος του 2018. Άρα η νομική ανάλυση της έκθεσης Όλαφ και οι απαντήσεις των Γκρικών αρχών θα πάρουν σε μάκρος ακόμα. Αυτό δεν είναι θετικό, ομολογουμένως. Από την άλλη, ενδεχομένως να μην αποτελεί μεγάλο πρόβλημα, γιατί έχουμε ακόμα 5% των πόρων μέχρι την ολοκλήρωση των υποθέσεων αυτών. Υπάρχει λοιπόν περιθώριο διόρθωσης με το 5%. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επιλογή των ε, προγραμμάτων, τελευταίο σημείο. Mm. Όπως είπατε, αυτό αποτελεί καθήκον των εθνικών αρχών. Και για τις δύο προγραμματικές περιόδους, και για την παλιά και για την καινούρια, οι διαδικασίες επιλογής ήταν εμφανείς, τις οποίες ε, και εν μέρη παρακολουθήσαμε. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε, θέλετε, με μονομένα ζητήματα και προφανώς είμαστε διευθυμένοι να σας βοηθήσουμε, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να λάβουμε και πολλές απαντήσεις από ογκρικής πλευράς για να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματά μας. Ε, Μακρηγόρησα. Ναι, να πάρετε το λόγο κι εσείς από τον τομέα ε, του ελέγχου, παρακαλώ, συνάδελφό σας. Ναι, ευχαριστώ. Θέλω να συμπληρώσω μερικά πράγματα. για τα όσα κάνουμε στην Ουγγαρία, σύστημα διαχείρισης και ελέγχου βλέπουμε ότι είναι αρκετά στεναρό. Εάν σημειωθούν αδυναμίες, προχωρούμε σε διορθωτικά μέτρα. Σωστά επισημαίνει ο Τόμας ότι στην ελεκτική δραστηριότητα είχαμε ζητήματα στις δημόσιες προμήθειες. Και γι' αυτό είναι πιο υψηλό το επίπεδο και για την Ουγγαρία των διορθώσεων για το 12-13. 14 με 20 ενισχύουμε το πλαίσιο διαβεβαίωσης, δεν περιοριζόμαστε στο 10% δηλαδή. Μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου περιμένουμε τη λογοδοσία και βέβαια έχουμε ξεκινήσει δουλειά ελεγκτική για τις δημόσιες προμήθειες και τις επιλογές. Προχωρούμε και μετά την ελεγκτική δουλειά που έχει γίνει μπορούμε να πούμε ότι πώς πραγματοποιήθηκαν από τις αρχές σημαντικές διορθώσεις ε, στο σύστημα. Ε, αυτά έχω να προσθέσω για το κλείσιμο. Όντως δεν μπορούμε να κλείσουμε τα προγράμματα στην Ουγγαρία. Έχουμε το 5% ακόμη των κονδυλίων που έχουν παρακρατηθεί μέχρι ότου διευθετηθούν όλα τα ζητήματα και δεν νομίζω ότι θα εκταμιευθούν αυτά τα κονδύλια προς το παρόν. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Άρα βλέπουμε ότι κάνετε καλή δουλειά. Γίνεται καλή δουλειά και οι Ουγγρικές αρχές, όπως βλέπουμε, είναι διατεθειμένες να αναλάβουν αυτές τις δραστηριότητες, να προχωρήσουν σε διάλογο. Κύριος Ίγκλε μας ε, το θύμισε ότι και ο Άγιος φοβέρα φέρει. Άρα λοιπόν καλά προχωρούμε μέχρι να λυθούν όλα τα ζητήματα. Θα συνεχίσουμε. Αν δεν έχει κανείς άλλο ζητήσει το λόγο, ο κύριος Ντόιτς και ο κύριος Γιάμετα. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να κάνω κάποιες ε, σύντομες παρατηρήσεις. Καθώς ήμουν μέλος της αντιπροσωπείας, εκτός ποσοστώσεως, με το ΣΥΠΗΝ, ως προερχόμενος από τη χώρα βουλευτής έλαβα μέρος στην αποστολή αυτή στην Ουγγαρία. Τρία πράγματα θέλω να πω. Η πρόεδρος λοιπόν εκπώνησε έκθεση στην οποία βλέπουμε πως είχε τρεις στόχους η αποστολή. Γιατί είχαμε ήδη πάει το 2011 στην Ουγγαρία. Θέλαμε να κάνουμε λοιπόν το follow-up, να δούμε τις εξελίξεις μεταξύ, Μετά τους στόχους του 2020, σε ποιο βαθμό έχουν υλοποιηθεί. Περιφερειακή ανάπτυξη και επενδύσεις από το 2014 μέχρι το 2020. Ε, πώς απορροφώνται, σε τι προσφέρουν ε, στην επίλυση των προβλημάτων αυτά τα κονδύλια, δηλαδή στη συνοχή και το καθεξής. Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας επίσης, το οποίο έχει την έδρα του στην Βουδαπέστη, και είδαμε μια ε, ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου που αφορούσε ακριβώς το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας. Για τους δύο πρώτους στόχους. Πολύ σύντομα. Βλέπω κάποιες ελλείψεις στις δύο πρώτες εκθέσεις, στους δύο πρώτους στόχους. που επιβεώνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις ε, τοποθετήσεις της. Σε σχέση με το follow-up ε, δεν βλέπουμε τίποτα μέσα στην έκθεση. Εμείς λοιπόν πήγαμε το 2011 στην Ουγγαρία, είδαμε τι ε, χρήματα διατίθενται από το Περιφερειακό Ταμείο και μετά το 2017 επισκεφθήκαμε και πάλι την Ουγγαρία για να δούμε πώς έχει προχωρήσει η κατάσταση, τι τάσεις υπάρχουν, θετικές, αρνητικές, στασιμότητα. Η προγραμματική περίοδος 7-13 είναι διαφορετική από αυτήν της περίοδου 14-20. Ε, ένα λεπτό όμω, ο κύριο από την Επιτροπή μίλησε 7-10 λεπτά. Είναι σημαντικό βέβαια το θέμα, όσο και αν ε, πρέπει να μιλήσουμε λίγο παραπάνω. Αν διαβάσει λοιπόν κανεί αυτήν την έκθεση, βλέπουμε ότι, υπογραμ... ότι δεν υπογραμμίζει τις προσωπικές εντυπώσεις που είχαμε ε, αποκομίσει εμείς από την επίσκεψη αυτή στην Ουγγαρία. Είναι φιλοευρωπαϊκό κράτος, ε, πραγματοποιεί επενδύσεις με συγχρηματοδότηση, εθνικά κονδύλια, ευρωπαϊκά κονδύλια, έχει αυξηθεί η απασχόληση, είναι πολύ χαμηλή η ανεργία. Η ανάπτυξη κινείται σε ποσοστά άνω του 4%. Η μισθή επίσης ε, αυξάνονται διαρκώς Βεβαίω δεν είναι η γη της επαγγελία, αλλά μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι υπάρχουν κάποια θετικά στην έκθεση αναφέρεται ότι είναι πολύ σημαντικό να καταγράφονται τα ποσά και σημειώνει τα σημαντικά ποσά τα οποία πηγαίνουν στην Ουγγαρία κτλ. Αλλά, αλλά δεν είναι αυτό η ουσία. Και αυτό που θέλω να πω ουσιαστικά είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη κάνει τις δηλώσεις τις οποίες βλέπουμε να επαναλαμβάνονται μέσα στην έκθεση. Έχει τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβεί στις συγκεκριμένε αναλύσεις. Έχει κάνει τη δουλειά της, έχει καταλήξει κάποια αποτελέσματα, έχει επιβεβαιώσει τη δουλειά στην Ουγγαρία. Και αυτό βλέπουμε να επανέρχεται μέσα στην έκθεση. Χωρίς καν κάποια παραπομπή σε πηγές. Πιστεύω ότι πρέπει αυτές οι αποστολές ε, στις χώρες πρέπει να έχουν ένα προσθέμενο, μια προσθέμενη αξία. Τι νόημα έχει να δίνουμε τόσα χρήματα για να πάμε στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Ουγγαρία. Όταν θα μπορούσαμε ωραιότατα να έχουμε μείνει στις Βρυξέλλες να στηριχθούμε στις μελέτες των υπηρεσιών μελετών του Κοινοβουλίου και να καταλήξουμε πάλι στην ίδια έκθεση. Δεν βλέπω κάτι το πρόσθετο δηλαδή να μας προσφέρει αυτή η έκθεση. Μόνο σε μια δύο Για τις ε, δημόσιες προμηθείς του αγωνισμούς με ένα μόνο πλειοδοτούντα. Με έναν μόνο μάλλον υποψήφιο λέγεται ότι υπάρχουν κάποιοι δημόσιοι διαγωνισμοί που έχουν μόνο έναν ε, υποψήφιο. Ένα λεπτό όμω αυτό αντιστοιχεί σε ένα, 24% για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ο αντίστοιχο μέσο όρο. Δεν είναι ότι κανένα κράτο στην Ένωση δεν έχει ε, καμία ε, διαδικασία με ένα μόνο υποψήφιο. Επομένω, ο μέσο όρο ευρωπαϊκό είναι 24%. Εντάξει, εμά είναι 36%. Και αν κοιτάξουμε και τα κράτη τα νεότερα κράτη-μέλη, δηλαδή εκείνα που μπήκαν το 2004, όχι Γερμανία, Γαλλία, κράτη Μπενελούξ, παλαιότερα κράτη, αλλά τα νεότερα κράτη-μέλη, τότε η Πολωνία 26%, η Τσεχία 41%, η Κύπρος, η Ρουμανία 38%. Αντίστοιχα ποσοστά διαπιστώνουμε. Είναι τόσο πολύ το 38% συγκρινόμενο με τα ποσοστά αυτών των κρατών. Γιατί νομίζω δεν προσφέρει τίποτα να δίνουμε στοιχεία χωρίς κάποιο μέτρο σύγκρισης, χωρίς να είμαστε υπερήφανοι για αυτό το 36%. Δεν μπορεί κανείς να μας κατηγορήσει το, το χειρότερο ή ότι είναι πάρα πολύ κακό το αποτέλεσμα αυτό. Επομένως, Λέτε στην έκθεση ότι η Επιτροπή θέλει, η Επιτροπή Κόντ ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασχοληθεί ειδικά με την Ουγγαρία κτλ. Δεν είναι κάτι το οποίο εμείς έχουμε εγκρίνει ως πρόταση. Δεν ξέρω αν είναι γνώμη της ε, Προέδρου μόνο, αλλά πάντως μου φαίνεται κάπως παράξενα παρουσιάζεται ως ε, θέση της Επιτροπής μας. Και σημειώνω ότι είναι δύσκολο να διασκεδαστεί η υποψία πως ε, μπορεί πάλι να ανοίγει μία διαδικασία εξεταστική, να μπει δηλαδή η Ουγγαρία στο εδόλιο, που ίσως αυτό να έχει και κάποια σχέση με την μεταναστευτική πολιτική, γιατί είναι άσχετα τα θέματα αυτά, δεν πρέπει να συμβεί κάτι τέτοιο. Άλλο είναι τα περιφερειακά κονδύλια και άλλο είναι η παροχή υποστήριξης ε, κάποιων κρατών ή μάλλον η μη παροχή υποστήριξης κάποιων κρατών στην πολιτική για τους ε, μετανάστες που έχει χαράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρω ότι η Επιτροπή αυτά τα αναμειγνιασμένος. Αλλά νομίζω ότι αν θέλουμε να επικρίνουμε κάτι σχετικό με την πολιτική μετανάστευση, το κάνουμε. Βεβαίω. Κανένα πρόβλημα. Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Αλλά ας μην δίνεται και η εντύπωση ότι ε, η πρόταση για περαιτέρω διερεύνηση και τα λοιπά εδώ εξυπηρετεί την ε, πίεση, το στόχο του να ασκηθεί πίεση στην Ουγγαρία για τη μεταναστευτική πολιτική. Μπορεί, μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θελήσει να κάνει έρευνες, Μπορεί να χρειάζεται, να είναι χρήσιμο κάτι τέτοιο στις συζητήσεις που είχαμε κάνει για το κράτος δικαίου, όταν είχε γίνει η συζήτηση για το κράτος δικαίου στην Ουγγαρία, είχε κάνει δεκτή αυτή η πρόταση η Επιτροπή, είχε μιλήσει για ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. για μια ενιαία μεθοδολογία με βάση την οποία θα πρέπει να εξετάσει την κατάσταση σε όλα τα κράτη. Και αυτή η ενιαία μεθοδολογία λοιπόν εφαρμοζόμενη στην Ουγγαρία δεν έδωσε αποτελέσματα δυσμενή αρνητικά για το κράτος δικαίου. Μπήκαμε στον κατάλογο του ενός, στο οποίο συμπεριλαμβανόταν και το ένα τρίτο των λοιπόν κρατών. Άρα λοιπόν θέλετε παραπάνω εξέταση, αναλύσεις και τα πολύ καλά, πολύ ευχαριστώ. Αλλά να συγκρίνουμε και με τα άλλα κράτη, να είναι συγκρίσιμα ενιαία μέθοδο, ενιαίε προϋποθέσεις, συνθήκες, όροι. Με χρονοδιάγραμμα ενιαίο που θα ισχύει και για τα 28 κράτη-μέλη, με εκθέσεις ανακράτος, γιατί κανένα κράτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι άμυρο αυτών των ε, ταμείων. Ε, όλοι, όλοι δηλαδή παίρνουν, όλα τα κράτη παίρνουν, ακόμα και οι καθαροί δωρητές ε, έχουν ε, τέτοια προγράμματα. Και τα κράτη δωρητές δηλαδή. Η Πρόεδρος, κοιτάξτε σας πω, για παιδιαρίσματα δεν έχω όρεξη ούτε χρόνο. Για τα, ε, τις διάφορες συναντήσεις που είχαμε, και δεν τα μασάω εγώ αυτά, δεν ήσουν παρόν όταν γινόταν η προετοιμασία. Κάνουμε μια προσπάθεια, το έχουμε πει αυτό για την Ουγγαρία ιδιαίτερα, γιατί είναι σημαντικό κράτος μέλος, θέλουμε να προχωρήσει, δεν θέλουμε να μείνει πίσω. Με έχει καθυβρήσει η κυβέρνηση της Ουγγαρίας, φτάνει τώρα όμως. Ο κύριος Γιάβου, έχει το λόγο. <clears throat> Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι λίγο πιο σύντομο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γραμματεία για την έκθεση. Είναι σωστή, εντελεχής και ακριβής. Και αποτυπώνει αυτά που είδαμε και διαπιστώσαμε. Έχω κάποιες ερωτήσεις και κάποιες λίγες προτερήσεις. Η κυρία Πρόεδρος είπε μόλις ότι ακόμα περιμένουμε κάποιες πληροφορίες σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα της πόλης της Βουδαπέστης. Δεν μας έχουν χορηγήσει πληροφορίες σε ό,τι αφορά την επιλογή των προγραμμάτων επίσης. Εξακολουθούμε να έχουμε αντιευκρίνηστα τα ζητήματα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις ελλείψεις αυτές που διαπιστώνουμε, θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον θα περιμένουμε περαιτέρω για τις πληροφορίες αυτές και μόνο όταν τις λάβουμε, θα ολοκληρώσουμε την έκθεση ή κατά πόσον θα ολοκληρώσουμε στο σημείο αυτό την έκθεση και θα περιμένουμε ακόμα εκ των υστέρων τις πληροφορίες ε, από την Ουγγαρία. Δεύτερη παρατηρήση όπως είπε και ο συνάδελφος, σε ό,τι αφορά τον έλεγχο από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το θέμα στην προκειμένη περίπτωση είναι τα λειτουργικά προγράμματα σε πρώτο επίπεδο. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλετε να υπάρχουν σαφείς ε, στόχοι. Από πλευράς της όλα φερευνώνται μεμονωμένα προγράμματα, τα οποία όμως ε, δειγματοληπτικά ε, επιλέγονται. Δεν είναι συστηματικός ο έλεγχος. Έχω μία έκθεση της Όλαφ του 2016 που δεν επισημαίνει τα προβλήματα τόσο πολύ στο λειτουργικό σκέλος, αλλά μάλλον στο θέμα της ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων και πώς οργανώνονται. Εδώ λοιπόν υπάρχουν περιπτώσεις ε, όπου υποπτευόμαστε ότι ενδεχομένω να υπάρχει διαφθορά και όλα αυτά έκανε τεκμεταλλοπτικούς ελέγχου. οι οποίοι είχαν, ε, εντόπισαν άμεσα προβλήματα. Περίπου 4% των δημοσίων συμβάσεων θα πρέπει να επιστραφούν στο πλαίσιο τη της διόρθωσης. Το οποίο για δειγματρεπτικούς ελέγχους είναι πολύ ψηλό ποσοστός και ο πραγματικός κίνδυνος είναι κατά πόσον υπάρχει καν μηχανισμός ελέγχου που ελέγχει το πλαίσιο των λειτουργικών προγραμμάτων και κατά πόσον συνάδουν με τις ε, ευρωπαϊκές άρχες ε, για τις δημόσιες συμβάσεις και συστηματική διαφθορά κατά πόσο έχουν διευκρινιστεί αυτές οι αιτιάσει για διαφθορά. Δεν υπάρχει λοιπόν τέτοιο συγκεκριμένο έλεγχο. Αν δεν γίνουν λοιπόν αυτοί οι έλεγχοι, τα προβλήματα δεν θα επιληθούν. Δεν θα αντιμετωπιστούν τα συγκεκριμένα σημεία κριτική κατά πόσον ε, δαπανήθηκαν σωστά τα ευρωπαϊκή πόροι κτλ. Κατά πόσον ε, εξυπηρετούν ε, δημόσια ιδιωτικά συμφέροντα. Μία ερώτηση έχω να κάνω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην έκθεση μιλάμε για την περίοδο 2014-2020. Η Ουγγρική κυβέρνηση θέλει να καλύψει την περίοδο αυτή με συμβάσει έργων. Αν συμβούν όλα αυτά τόσο γρήγορα, το 2018 λοιπόν, μετά τις εκλογές του Απριλίου, η καινούργια κυβέρνηση δεν θα έχει ελευθερία διάθεση ε, των ε, μέσων αυτών. Η σημερινή κυβέρνηση θέλει να δαπανίσει όλα τα υπόλοιπα αυτά μέσα, όλα αυτά τα υπόλοιπα κονδύλια, όπως ε, θεωρεί σωστό. Για την περίοδο μέχρι το 2020 ο κίνδυνος λοιπόν είναι επί δύο-τρία χρόνια να μην ε, κατατεθούν οποιαδήποτε, οποιασδήποτε νέες ιδέες και όλα να ακολουθήσουν ε, την παλιά, το πατημένη, το παλιό αυτό σχέδιο και αυτό να οδηγήσει σε οικονομική, δημοσιονομική αστάθεια. Ευχαριστώ. Να πω στον συνάδελφο Γιάβορο ότι στο πρόγραμμα Heart of Budapest καλό θα ήταν... Έχουμε τα τεκμήρια από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό που μας λείπει είναι οι γνωματοτήσεις της εγκουρικής κυβέρνησης και γι' αυτό λοιπόν καλό θα ήταν να είχαμε όλη την ανταλλαγή αυτών των επιστολών για να διαπιστώσουμε ακριβώς τι αφορούσε η συζήτηση. Άρα θέλουμε, Τόμας, και την ουγγρική αλληλογραφία, γιατί αυτό θα επηρεάσει και το πώς εξετάζουμε την έκθεση της όλα, που δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτή τη στιγμή, γιατί μας λείπουν πληροφορίες. Αυτό που μας λείπει είναι επίσης οι πληροφορίες από την ε, εισαγγελία για το μετρό, την ε, γραμμή 4. Περιμένουμε λοιπόν ε, τις απαντήσεις αυτές. Αν υπάρχει κάποια τροπολογία να την καταθέσετε, αλλά επί του προεχόμενου μας λείπουν διάφορα στοιχεία. Αλλά σε γενικές γραμμές αυτές οι εκθέσεις δεν παροβάλλουν πληροφορίες. Στον κύριο Μπέντε και την κυρία Άρανοφ να δώσουμε το λόγο για να απαντήσουν τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Μια ερώτηση έχω σημειώσει από τον κύριο Γιάβορα, αν καταλαβαίνω καλά, για την ταχεία υλοποίηση. Είναι δίκοπο μαχαίρι. Ξέρετε ότι συνολικά στα κράτη-μέλη είναι κάπως πιο αργή η πρόοδος στην αρχή της προγραμματικής περίοδου και χαιρόμαστε ιδιαίτερως για το ότι οι Ουγγρικές αλλά και άλλα κράτη-μέλη και οι Ουγγρικές Αρχές όμως έχουν επιταχύνει κάπως ε, τις ε, διαδικασίες υλοποίησης. Από την άλλη βεβαίως ε, πρέπει να συζητήσουμε, έχουμε συζητήσει κάποια προβλήματα, εκ των οποίων ορισμένα τα καλύψατε ήδη. επί παραδείγματι ότι δεν υπάρχει αποθεματικό για πιθανές περαιτέρω κρίσεις απρόβλεπτες αυτή τη στιγμή. Μέχρι την προσεχή προγραμματική περίοδο δεν υπάρχουν τα κονδύλια όπως επίσης ότι μαζεύονται όλα, όλες οι διαδικασίες ε, ε, εκδήλωση ενδιαφέροντος και προκηρύξεις, ε, διαγωνισμοί στην ίδια περίοδο με υπερβολική επιβάρυνση και στην πρακτική σκόπια και ταυτόχρονα στην εξέλιξή τους. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με την ε, παράλληλη εξέλιξη του ερωτικού και του, και του κοινωνικού ταμείου. Πρόκειται για μια επιβάρυνση υπερβολική μέσα σε ένα έτος. Από την άλλη όμως βλέπουμε με ικανοποίηση ότι ε, προχωρούν ε, οι εκταμιεύσεις ομαλά και μάλιστα βαίνουν τα χρήματα προς επενδύσεις στις κοινότητες, στις περιφέρειες κτλ. Περισσότερα δεν έχω να σας πω αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ ε, για τα ε, ποσοστά αυτά για τους Ε, για ένα μόνο, με ένα μόνο ενδιαφερόμενο έχουμε την Κροατία και την Πολωνία με 55% και μετά ακολουθεί η Ουγγαρία με 36%. Εντάξει, ε, επομένως δεν είναι και τόσο καλά τα αποτελέσματα και πρέπει να δούμε βεβαίως γιατί ειδικά αυτές οι τρεις χώρες. Η Γενική Διεύθυνση μπορεί να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Για τη Γενική Διεύθυνση για τον πολιτισμό ίσως πολύ πολύ σύντομα αν θέλετε γιατί έχουμε και άλλο ένα θέμα στην ημερήσια διάταξή μας. Παρακαλώ. Έτσι είχα εγώ τουλάχιστον σημειώσει μπεγκόνια. Αράνο, εσείς είσαστε γυναίκα ή κάνω λάθος. Ε, δύο λεπτά από το πολύ όμως. Χωρίς μικρόφωνο. Ε, I will be very, very... Α, είμαι πολύ σύντομη. Γιατί εμείς Κάνουμε αυτή την ε, αποστολή, την επίσκεψη του Ευρωπαϊκού Ίδρυμα Τεχνολογίας και από ό,τι κατάλαβα από την έκθεση είχαμε κάποια θέματα τα οποία αναλύθηκαν, τα οποία αναδείχθηκαν από την συζήτηση με τον Διευθυντή ε, που μίλησε στον δικό μας Διευθυντή και από ό,τι καταλάβαμε Τα θέματα τα οποία εκκρεμούν και αναδύθηκαν ήταν όσο αφορά τις ανοιχτές δράσεις είναι αυτές που επισήμανε στην έκθεση του του Ελληνικού Συνέδριου. Αλλά να σας εξηγήσω με λίγα λόγια το ότι έχει αναλυθεί δράση για αυτά τα θέματα που ακόμα εκκρεμούν. Το είναι των ανοιχτών δράσεων όσον αφορά την ε, τροποποίηση του κανονισμού. Βρίσκεται να εξελίξει το θέμα, ασχολούμεθα τώρα με μια σειρά τροποποιήσεων που δεν θα έχουν επιπτώσει στο ε, επόμενο ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Οπότε έχουμε αυτό το 25% της χρηματοδότηση που θα το αντιμετωπίσουμε στην ε, επόμενη τροποποίηση του κανονισμού. Επίσης, όσον αφορά το αν είναι εφικτά αυτά τα χρήματα που θα διατεθούν και επίσης να ληφθούν υπόψη αυτές οι τροποποίησεις στο επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο. Τώρα, στο ισχύον πρόγραμμα πλαίσιο και στο ορίζον 2020 δεν μπορούν αυτά να ενταχθούν. Όσον αφορά την εθνική αυτονομία, λήφθη η σχετική απόφαση και με την ευκαιρία να σας ανακοινώσω την πλήρη χρηματοοικονομική ανεξαρτησία για την πρώτη πρώτου του 18. Τώρα όσον αφορά το θέμα του προσωπικού προβλέπονται επιπλέον ανθρώπινοι πόροι όπως ζητήθηκε. Είπατε για την αύξηση στα 65 άτομα και σύμφωνα με το σχέδιο για το 2018 θα πάμε στους 68 προσωπικό. Θα ακούσουμε φυσικά το τι χρειάζεται το Ίδρυμα. Είπαμε ότι υπάρχει ένα άνω όριο 70 όσον αφορά το προσωπικό, αλλά και αυτό επιδέχεται ζήτηση στο μέλλον. Και εδώ βάζουμε τη λία προς το παρόν. Σας ευχαριστώ. Έχουμε ένα ακόμα... Ολοκληρώθηκε μάλλον το θέμα αυτό και να περάσουμε στο τελευταίο θέμα της ημερήσιας τατάξης. Μια πολύ ε, σημαντική ε, περίπτωση Rapid Case, νέο εργαλείο του Ρεκτικού Συνεδρίου για την ε, μείωση κατά 5% του προσωπικού στα ευρωπαϊκά όργανα. Ο κ. Ρούσο είναι ο εισηγητής, ο κ. Ashworth είναι ο δικός μας εισηγητής. Λυπάμαι για την καθυστέρηση, έχετε το λόγο κύριε Ρούσο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα αυτή τη άμεση επανεξέταση του ζητήματο για τη μείωση κατά 5% του προσωπικού. Έχω κάποιες διαφάνειες που μπορούμε να σας δείξουμε και νομίζω ότι έτσι θα είναι πιο σαφή μερικά σημεία. Τώρα θα σας πούμε. Μας ζήτησε το Συμβούλιο να κάνουμε μια τέτοια ανεξάρτητη ε, μελέτη ω προ την μείωση του προσωπικού κατά 5% όπως προβλέπει η Διοργανική Συμφωνία του 2013 και αυτό προβλέπει αυτή την βαθμία μείωση κατά 5%. Επί τη βάση αυτού, επομένως, προέβημε σε αυτή την επανεξέταση. Μπορείτε τώρα να δείτε τι προβλέπει αυτή η συμφωνία. Και θέλαμε να εξισορροπήσουμε την αύξηση του χρόνου εργασίας στις 40 ώρες εβδομαδίας. Όπως προβλέπει η απόφαση Κομισιόν και Συμβουλίου για το 5% σύμφωνα με το πρόγραμμα της πρώτης πρώτη του 2013. Αυτό αφορά όλους τους εργαζομένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως αυτή η μείωση ισχύει για όλα τα θεσμικά όργανα και υπηρεσίες. Αποφάσισε το Ελληνικό Συνέδριο να τα κάνει όλα αυτά στα πλαίσια της άμεξης επανεξέταση του ζητήματος, τόσο ώστε να αξιοποιήσουμε τις τελευταίες πληροφορίες και όλοι οι συναρμόδιοι να μπορούν να έχουν ταχεία ενημέρωση. Οπότε και θέλαμε εγκαίρως να ανακοινώσουμε τα σχετικά για να καλυφθεί η απόφασή μας από τη χρήση του οικονομικού έτους 16. Τώρα έχουμε τις εξής ε, χρονικές περιόδους ε, για αυτή μας την αξιολόγηση, κάνουμε τη διάκριση τώρα, όπως βλέπετε στις διαφάνειες. Αναφέρει η έκθεση τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους. 2013 μέχρι το 2017 αναφοράς σύμφωνα με τη Διοργανική Συμφωνία. Σε αυτή την περίοδο η μίσου του 5% πρόκειται βαθμιαίως να υλοποιηθεί. Δεύτερη περίοδος, 2012-2017. Είναι η περίοδος από τη μέρα που άρχισε να ισχύει το πρόγραμμα της μειώσεως του 5% μέχρι το έτος που θα γινόταν η πλήρης υλοποίηση της αποφάσεως. Τρίτη περίοδος, 2012-2016, πρόκειται για την περίοδο από την θέση σε ισχύ αυτού του προγράμματος μείωσης μέχρι το τελευταίο έτος για το οποίο τα στοιχεία για πραγματικές καταβολές και αποζημιώσεις θα ήταν έγκυκανο από την επανεξέταση. Βλέπουμε τώρα τι έγινε. Οι περισσότερες υπηρεσίες ε, υλοποίησαν αυτό το 5% όπως αποφασίστηκε από το σχετικό πρόγραμμα και μερικές καθυστέρησαν και από ένα σύνολο 2.306 θέσεων υπαλλήλων ε, που αποφασιζόταν πήγαμε στους 2.145 θέσεων που μειώσαμε και άρα υπάρχει ακόμα εστέρηση κατά 163 θέσεις που προβλέπεται να υλοποιηθεί μεταξύ 18 και 20 όπως τα δείχνει η διαφάνεια. Οφείλεται αυτή η καθυστέρηση το ότι η υπηρεσία εξωτερική υπηρεσία ήθελε να. Δεν κατάφερε μάλλον να ολοκληρώσει ε, το θέμα αυτό το, μέχρι το 2018 αλλά και κάποιες άλλες υπηρεσίε. Το Συμβούλιο αποφάσισε να ολοκληρώσουν εκτελεστικές υπηρεσίες μέχρι το 2020 και είναι σημαντικό να σας αναφέρω για όλα αυτά ότι οι περισσότερες μειώσεις θέσεων έγιναν με κατάργηση θέσεων που εχείρευσαν λόγω συντάξεως ή ασθενείας. Και θα επανέλθουμε σε αυτό σε λίγο. Έχουμε μόνο σε αυτή την ε, μείωση των θέσεων Έχουμε πάντως για την Κροατία 322 θέσεις που θεσπίστηκαν και κάποιες άλλες προσθήκες. Ας πούμε με την αλλαγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αλλά και στο Κοινοβούλιο. Πάντως, ακόμα και με αυτήν την αύξηση αυτές οι νέες θέσεις δόθηκαν σε εκτελεστικές υπηρεσίες και αποκεντρωμένες. Και σε αυτό θα επανέλθουμε. Κατά την λόγο περίοδο η Διευθυντική Αρχή αποφάσισε αυτό και έτσι επηρεάστηκε το σύνολο των θέσεων εργασίας. Όπως προέβλεπε το αρχικό σχέδιο. Βλέπετε τώρα πώς έγινε η εξέλιξη. Βλέπουμε τώρα η συνολική μείωση, σύμφωνα με αυτό το πρόγραμμα, ήταν το 1,1% το τελικό αποτέλεσμα. Αλλά έχουμε αυτό το μεσόρος έχουμε ως ε, διακύμανση μεταξύ της κάθε υπηρεσίας. Πάμε στο 3,5% μέσο όρο. Η αποκέντρωση στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες ήταν 13,7% και 42,9% στις ε, εκτελεστικές υπηρεσίες. Η διαφορά αυτού του 5% που αποφασίστηκε και τι έγινε στην πραγματικότητα και πρόκειται για το 1,1% είναι το ότι έχουμε κάποιες νέες θέσεις λόγω της προσχώρησης της Κροατίας. Όπως προείπαμε. Επίσης είχαμε μεταφραστές των Κελτικών για την Ιρλανδία. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης ε, είχαμε κάποιους υπαλλήλους πολιτικών ομάδων. Και επίσης έχουμε και κάποιες θέσεις που δόθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, για κάποιες νέες πολιτικές όπως ας πούμε την πολιτική μετανάστευση. Για να δούμε τώρα πώς είναι η θέση απασχόλησης. Είναι 0,4% για πρώτη πρώτη του 2013 μεχρι πρώτη πρώτη του 2017. Είναι θέσεις που πραγματικά κατέχονται από υπαλλήλου. Επίσης όπως προβλέπει το αρχικό πρόγραμμα έχουμε την μείωση των θέσεων όπως σας προανέφερα και η μείωση είναι κατά 1,3% και η αύξηση είναι 9,6% και 33,7% για τις κεντρικές υπηρεσίες, για τις απογειωμένες υπηρεσίες και τις ε, εκτελεστικές υπηρεσίες όπως βλέπετε. Και ταυτόχρονα οι θέσεις που χειρεύουν έχουν πέσει σημαντικά γιατί ακριβώς είχαμε την κατάργηση κάποιων θέσεων γιατί ακριβώς καταργήσαμε θέσεις που ήδη εχείρευαν ή που εχείρευσαν κατά την οικονομική χρήση, το οικονομικό έτος όπου βρισκόταν εν εξελίξει αυτή μας η ε, εργασία. Τώρα, η εξέλιξη όσον αφορά το κόστος του προσωπικού στα θεσμικά όργανα. Είχαμε για επαλλήλους και προσθένους επαλλήλους 11,5% αύξηση και και 9,2% για πραγματικές πληρωμές. Αυτό είναι λόγω της τιμαριθμικής αιτήσεως προσαρμογής που αφορά όλο το προσωπικό και κάποιες αυξήσεις μισθολογής λόγω των προαγωγών. Πότε έχουμε αυτή την φυσιολογική αύξηση λόγω της φυσιολογικής μισθολογικής εξέλιξης γενικός και ατομικός. Βλέπετε σε αυτό το γράφημα πως έχει κατάσταση για τις εκτελεστικές υπηρεσίες και τις αποκεντρωμένες πληρωμές και κόστος προσωπικού ακριβώς όπως προείπαμε Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ισηγητά, σας ε, ευχαριστούμε στην την ευκαιρία να παρουσιάσουμε αυτή μας την επανεξέταση. Είμαστε στη διάθεσή σας. Πρόεδρος. Οι διερμήνες μας δώσαν ακόμα 10 λεπτά. Κύριε Ashworth. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι σημαντική έκθεση και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ρουσο και το ελεγκτικό συνέδριο για τη δουλειά τους. Ε, θα είμαι σύντομος. Καλά νέα της έκθεσης είναι ότι το ελεγκτικό συνέδριο διαπιστώνει ότι το 5% μείωση του προσωπικού έχει επιτευχθεί και τι με κάποιες καθυστερήσεις. Αυτά ήταν τα καλά νέα. Τα κακά νέα όμως, τις λεπτομέρειες και ειδικότερα αν ε, κοιτάξουμε ποιες είναι οι παρεκκλήσεις και εξαιρετικές περιστάσεις αύξησης προσωπικού, ο περιορισμός του προσωπικού έφτανε μόνο στο 1,1%. Τρεις λόγοι λοιπόν παρουσιάζονται για αυτή την απόκληση. Πρώτον, και απόλυτα αιτιολογημένο, ήταν ότι ε, χρειάστηκε να ενισχυθεί το οργανόγραμμα μιας σειράς υπηρεσιών και φορέων λόγω της ένταξης της Κροατίας, λόγω των αναγκών σε διερμηνία για τα Ιρλανδικά, ενίσχυση του προσωπικού ασφαλείας, του προσωπικού του δικαστηρίου κτλ. Ωστόσο, η συμφωνία για τον περιορισμό φαίνεται να έχει ε, αποκλείσει λίγο πολύ το κοινοβούλιο και έχουν προσληφθεί πολλά ακόμα πρόσωπα το τελευταίο διάστημα. Επίσης ενδιαφέρον είναι, μέχρι και ύποπτο μπορώ να πω, το ότι στην πενταετία της συμφωνίας καταγράφεται αύξηση 33,4% των συμβασιούχων. Επίσης είναι ενδιαφέρον το ότι το κόστος του δημοσιονομικού αυξάνεται κατά 6% για το προσωπικό μεν, αλλά οι πραγματικές πληρωμές φτάνουν στα 9,2% αύξηση. Και έχω κάποιες ερωτήσεις για το ελεγκτικό συνέδριο. Πρώτον, μπορεί το ελεγκτικό συνέδριο να μας πει εάν υπήρξε εξοικονόμηση πόρων χάρη στη μείωση κατά 5% ή μήπως το κόστος απλώς μετακυλίστηκε κάπου αλλού. Δεύτερον, εάν οι πολιτικές ομάδες είχαν συμπεριληφθεί στο στόχο του 5%. Το Κοινοβούλιο πιστεύετε ότι θα είχε τηρήσει τις δεσμεύσεις του και θα υπήρχε κάποια αύξηση, μάλλον ε, θέσεων πέραν του 1,1%. Τρίτον, το Ελληνικό συνέδριο πιστεύει ότι το 5% μείωσης προσωπικού ήταν μια προσπάθεια άξια λόγου. Ξέρω ότι ο Επίτροπος Έτσιγκερ όπως και η έκθεση για το πολιτισμό νομικό πλαίσιο του Κοινοβουλίου, σημειώνω ότι πρέπει να, είναι μόνο άπαξ αυτή η, αυτό το εγχείρημα, να μην επαναληφθεί δηλαδή η περίοδος αυτής της μείωσης. Και τέταρτον, πιστεύετε ότι ήταν καλό προαίρετος ο ορισμός του 5% για περιορισμό του προσωπικού. Και εγώ πιστεύω ότι, κοιτώντας έτσι προς τα πίσω, ότι υπήρχαν και κάποιες αναπάντεχες συνέπειες. Δηλαδή, οργανισμοί οι οποίοι χρειάστηκε να αναλάβουν νέα καθήκοντα ε, και δραστηριότητες αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες. Φερρυπίν, συνάδελφοι της Επιτροπής μας είδαν επανειλημμένως από το ελεγκτικό συνέδριο να μας λέει ότι είχε μεγάλη επιβάρυνση. Η υπηρεσία εξωτερικής δράσεως επίσης, την προηγούμενη εβδομάδα μόλις, όπου μας έλεγαν ότι δυσκολεύονταν να κάνουν τη δουλειά τους καλά λόγω της ελλείψεως προσωπικού. Επίσης θέλω να ρωτήσω, οι στόχοι μείωσης έχουν οδηγήσει σε μία πιο, και σε εμά αλλά και στα άλλα όργανα, σε μία πιο εφάνταστη και δημιουργική διαχείριση του προσωπικού των ανθρωπινών πόρων. Για να καταλήξω. Οι στόχοι μείωση έχουν οδηγήσει σε αρνητικέ συνέπειε ω προ κάποιε δράσει και λειτουργίε Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, είναι σαφέ ότι σε, κάποιου τομεί ο προσδιορισμό στόχων μείωσης οδήγησε σε μετακύληση των διαδικασιών ε, και των επιλογών διαχείριση του προσωπικού. Τρίτον, οι πολιτικές ομάδες καλό θα είναι να κοιτάξουν τα δικά τους επίπεδα στελέχωσης και να ε, τις απασχολήσει το ερώτημα γιατί κάθε φορά που υπάρχει μείωση για τα λοιπά όργανα αποκλείονται από αυτό το κανόνα της μείωσης οι πολιτικές ομάδες. Και εν τέλει, Πρόεδρε δεδομένου ότι τα συνολικά, η ο συνολικός όγκος του προσωπικού και το κόστος του προσωπικού που κατέχει θέσεις έχει παρουσιάσει αύξηση κατά 0,4% κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Θεωρώ ότι μπορεί να ήταν καλοπροαίρετο ο στόχος της μείωσης κατά 5%, αλλά εν την πράξη απεδείχθη όργανο φωνικό και αμβλή. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι τα είπατε όλα, τα καλύψατε. Όλα αυτά τα οποία και εμείς ε, διαβάζοντας αυτές τις προτάσεις είχαμε διαπιστώσει. Ο κύριος Ρούσο έχει, κάνει, έχει δείξει πως θέλει να κάνει μια ερώτηση. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Άσουερθ, εισηγητή. ο οποίος από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχει πλήρη κατανόηση του περιεχομένου του εγγράφου μας και απέδωσε πολύ πιστά το περιεχόμενο αυτό με ένα πολύ ενδιαφέρον ε, φάσμα, πρέπει να πω, πολύ πιστό φάσμα της δουλειάς μας πέραν του γεγονότος ότι δεν πρόκειται για μια πραγματική έκθεση δημοσιονομικού ελέγχου, αλλά για μια εντάχει επισκόπηση μια συγκεκριμένη περίπτωση, ο στόχος μας, ο στόχος του Ελληνικού Συνεδρίου δεν ήταν να δώσουμε γνωμοδότηση, αλλά κάποιες πληροφορίες, κάποια στοιχεία. Είτε δημοσιευμένα, είτε όχι, προς τους ενδιαφερομένους εν προκειμένου το Κοινοβούλιο για να δώσουμε στο μέγιστο δυνατόν πλήρη εικόνα του αντικειμένου αυτής της μελέτης. Ωστόσο, Κάποιες ε, σκέψεις ή σχόλια καθαρά πολιτικού χαρακτήρα δεν αρμόζουν στο ελεγκτικό συνέδριο. Και για να ξεκινήσω από το τέλος, όπως το τα λέγανε και οι φίλοι μας οι Γάλλοι, το ελεγκτικό συνέδριο εξετάζει με βάση τη σκοπιμότητα την, την ίδια αυτή την επιχείρηση μείωσης, δηλαδή εξετάζει εάν πρέπει ή μπορεί να επαναληφθεί αυτή, αυτό το επιχείρημα μείωσης κατά 5% του προσωπικού. Αυτή ήταν η θεώρηση. Εγώ θα προσπαθήσω να απαντήσω στην συγκεκριμένη ερώτηση του εισηγητού για την εξοικονόμηση πόρων. Είναι σαφές νομίζω το πόρισμα αυτών των ε, εκθέσεων μας, της έκθεσής μας. Η εξοικονόμηση πόρων δεν υπήρξε τουλάχιστον όχι άμεσα συνδεδεμένη με, την, ε, με τον περιορισμό του 5%, κατά 5% του προσωπικού μόνο στις αναλήψεις υποχρεώσεων και πραγματικές πληρωμές, δηλαδή στον προϋπολογισμό βλέπουμε να αντικατοπτρίζεται κάτι τέτοιο μόνο στα νούμερα του προϋπολογισμού. Ε, γιατί ναι μεν υπάρχει ένας υπολογισμός ποσών ο οποίος τελικά υπολείπεται αυτού που πραγματικά κατεβλήθη. Από την άλλη υπάρχουν και οι αυξήσεις των μισθών, ε, φυσιολογικές αυξήσεις, είτε πρόκειται για την τερμορυθμική αναπροσαρμογή, είτε πρόκειται για την ε, προσωπική πρόοδο του προσωπικού στη σταδιοδρομία του, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό προσωπικού, με, την, ε, με τις προαγωγές που οδηγούν και σε αύξηση μισθών, τότε βέβαια δεν έχουμε εξοικονόμηση πόρων. Και για να απαντήσω στην ερώτηση και για τις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το προσωπικό τους, όντως αυτές αποκλείστηκαν από τη συμφωνία και άρα δεν τις καλύπτει η έκθεσή μας. Και τα στοιχεία που σας παρουσιάσαμε. Σε σχέση με τη σκοπιμότητα του εγχειρήματο, όπως είπα, δεν πιστεύω ότι πρέπει το ελεκτικό συνέδριο ή ότι δικαιούται το ελεκτικό συνέδριο να τοποθετηθεί στο θέμα αυτό. το γεγονός ότι κάποια θεσμικά όργανα με συγκεκριμένα ή φορεί με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως το ε, δικαστήριο ή όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης αντιμετώπισαν δυσκολίες λειτουργίας λόγω υποστελέχωσης ίσως σε ένα βαθμό να ήταν αναπόφευκτο δεδομένης της μεγάλης ποικιλία και του ευρωαίου φάσματο αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των διαφορών φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή. Και χωρίς να βλέπω κάποια πρόθεση πίσω από αυτό, θα μπορούσε η λειτουργία των ευρωπαϊκών φορέων να έχει περιοριστεί με, αυτή την, ε, με αυτό το πρόγραμμα περιορισμού γιατί τουλάχιστον το πεδίο της συμφωνίας ήταν, είχε και σαν στόχο να αυξηθεί η παραγωγικότητα και να εξωτερηθεί ως εκ τούτου το κόστος της εργασίας με την αύξηση του χρόνου εργασίας του εβδομαδιαίου σε 40 ώρες. Αυτό, αυτό δεν έχει αλλάξει. Σας ευχαριστώ και έτσι ολοκληρώσαμε τη σημερινή συνεδρίαση. Κύριε Στεχόφτσκι, δεν έχουμε πλέον διερμηνία, γιατί μας έδωσαν 10 λεπτά παραπάνω διερμηνής. Ναι, αγγλικά αν θέλετε. Σας ευχαριστώ ευγενικά, η πρόεδρος σας ευχαριστώ, κύριε Μηνής και σας ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Thank you very much. I will be very briefly thanks interpreters for staying here. It was a long question of reporter. Thank you very much for your question. But my question is about that